Good morning, colleagues, um, and I'm going to begin, try and begin on time. I'm starting to... Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε εγκαίρως. Να μην ε, καθυστερήσουμε από το πρωί. Γιατί είναι άδικο για τους συναδέλφους που είναι πάντα στην ώρα τους. Λοιπόν, Είμαστε στο σημείο 19 για αρχή. Παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων 2013-2015, πρόγραμμα εργασίας 2016-2018, Κλάρα Κουέρα, από την πρόεδρο της ομάδας συντονισμού εποπτής του ΣΥΣ2. Εισαγωγικά λοιπόν να σας καλωσορίσω εφαρμογή των διατάξεων ε, για την ε, εποπτεία του συντονισμού του ΣΥΣ από πλευράς των εθνικών οργών είναι πολύ ε, σημαντική και κέρια αυτή η έκθεση. Η κυρία Γκουέρα θα μιλήσει και για την δουλειά που προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια. Χωρίς άλλοι σα σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε για να παρουσιάσω τις δραστηριότητε της Ομάδας Συντονισμού Εποπτείας του ΣΥΣ2. Είναι σημαντικό το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή σας θέλω ιδιαίτερος για μας για τα θέματα προστασίας των δεδομένων. Ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς που ζούμε τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, πολιτών. Η εποπτεία η ομάδα αυτής, αυτή εποπτείας συντονίζει τον εποπτικό μηχανισμό ε, για την επίβλεψη του συστήματος ε, Σέγγεν. Έχουμε εδώ και 20 χρόνια συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί αντικατοπτρίζει τη δομή του κανονισμού του 2006 και την απόφαση του 2007. Με το νέο αυτό νομικό πλαίσιο το ΣΥΣ ε, επέκτησε νέα στοιχεία και διαφορετικούς κανόνες συντονισμού μεταξύ των οποίων θέλω να υπογραμμίσω την εισαγωγή της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά τα στοιχεία των ανθρώπων. Είναι σημαντική η, των ατόμων, είναι σημαντική αυτή η διαφορά. Δεύτερον είναι να αιτιολογηθούν Οποτεδήποτε τα στοιχεία πρέπει να διατηρηθούν για μακρύτερε περιόδου και τέλο ε, η δημιουργία συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση των δικαιωμάτων των ε, ατόμων. Νέοι κανόνε για την προστασία λοιπόν των δεδομένων που είναι ευπρόσδεκτοι. Επίσης θεσπίστηκε ένα νέο μοντέλο εποπτείας με μια νέα δομή που περιλαμβάνει τις εθνικές αρχές και τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαίο επόπτη δεδομένων, το DPS. Ε, δηλαδή τους οργανισμούς προστασίας δεδομένων, τους εθνικούς και τον ευρωπαϊκό. Η ομάδα μας είναι καινούρια και χρειάστηκε να προβούμε σε επιλογές όσον αφορά τις ομάδες εργασίας μας. Είμαστε μια δομή που αποτελείται από 30 μέλη, συν τρεις παρατηρητές, οπότε προσπαθούμε να το έχουμε μια ευελιξία ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. προτάσουμε την ε, τα email με συγκεκριμένο δίκτυο για να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και φτιάχνουμε και ομάδες για να εξετάσουμε συγκεκριμένα θέματα πιο εις βάθος. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνεργασίες, συνέργειες με τις άλλες ομάδες εποπτείας για θέματα Σέγγεν όπως το FIS και το Eurodac. Υπάρχουν ομάδες και εκεί, υπάρχουν κάποια, υπάρχει και κάποια σύμπτωση στα μέλη, δηλαδή και έτσι προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και να αποφεύγουμε την επικάλυψη εργασίας καθώς και, τη, και, ε, επιδιώκουμε τη συνεργασία και όπου αυτό γίνεται. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω δύο βασικές ε, γραμμές Άξονε μάλλον. Πρώτον, έχουμε τα συγκεκριμένα θέματα που καθορίζονται από τα γεγονότα, από τις εθνικές ε, ε, αρχές προστασία δεδομένων ή θέματα που απαιτούν άμεση δράση. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και μάλιστα ήταν και το πρώτο μας, ήταν το επεισόδιο hacking της Δανία. Το 2013 ο Διευθυντής του Οργανισμού της Δανέζικης ε, Αρχής Προστασίας Δεδομένων ανέφερε αυτό το περιστατικό που ήταν τεράστια ρήξη ε, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και αυτή η ε, ρήξη αντιμετωπίστηκε εντό της Δανίας από τη Δανέζικη DPA και την παρακολούθησε και όλα στην εξέλιξη η Δανέζικη DPA μας παρουσίασε τα τελικά της πορίσματα δε πέρυσι για το, την έρευνα που έγινε τότε και επίσης το παρακολούθησε και η Κομισιόν και η ομάδα που δημιουργήθηκε με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ε, οι εθνικές αρχές προστασίας ε, δεδομένων δεν αναμίχθηκαν άμεσα. Αυτό ήταν κρίμα διότι αυτού του είδου η, παρα... ρήξη έχει αντίκτυπο σε όλα τα κρατημέλη και θέτει σε κίνδυνο τα στοιχεία όλων των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα προσπάθησε να συνδεθεί με τις δραστηριότητε που γίνονταν και καταφέραμε να είμαστε παρατηρητές στην ειδική ομάδα που δημιουργήθηκε. Συμβάλαμε λοιπόν σε εθνικό επίπεδο, προβήκαμε σε δράσεις, ενέργειες, ήρθαμε σε επαφή με τις εθνικές μας αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθεί το τι ακριβώς γινόταν για το περιστατικό αυτό και για το κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Και αυτό έγινε με πολύ συντονισμένο τρόπο. Αυτό ήταν ένα θέμα λοιπόν που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν μια πρεμιέρα για την ομάδα μας και δεν... Ε, ε και το παρακολουθήσαμε για δύο χρόνια, αλλά δεν έχουμε πια πληροφορίες, δεν ξέρουμε δηλαδή το εύρος της παράβασης, της ρήξης. Κάτι ε, ακόμα που μας ζητήθηκε είναι να δώσουμε ερμηνεία του νομικού πλαισίου, όποτε υπάρχουν νομικά προβλήματα να προσπαθούμε να βρούμε κοινέ λύσεις. Οπότε δώσαμε έτσι και τη γνώμη μας για ε, συστηματική αντιστήχηση και, και διασταύρωση πληροφοριών για τα σύνολα των πληροφοριών. Η γνώμη μας ήταν αρνητική για, ότι δηλαδή αυτό δεν ανέπεπτε, δεν εντασσόταν μάλλον στο νομικό πλαίσιο. Είπαμε ότι οι αρχές δεν θα έπρεπε λοιπόν να το κάνουν, γιατί αυτό ε, ήταν η παράβαση της αρχής περι, περιορισμού του στόχου. Η Europol επίσης έχει φτιάξει ένα νέο σύστημα ελέγχου, πράγμα που σημαίνει ότι η Europol έχει στόχο να μπει μέσα σε όσου έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΣΥΣ. Το αναλύσαμε κατά πόσο αυτό ήταν δυνατόν. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση γι' αυτό, αλλά αυτό αφορά και την ίδια τη Europol. Ένας άλλος άξονας είναι πιο διαθροτικός πιο δομικό, δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα ζητήματα όπως αυτά προκύπτουν, αλλά επενδύουμε σε πιο μακροπρόθεσμη εργασία. Αυτό κάνουμε και αυτή ήταν μια βασική δραστηριότητα που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, να αναπτύξουμε δηλαδή ένα κοινό πλαίσιο ε, ελέγχου. Όπως γνωρίζετε, το νομικό πλαίσιο για το ΣΥΣ απαιτεί από τις αρχές ε, προστασίας ε, δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διενεργούν έλεγχο με βάση ε, συγκεκριμένα πρότυπα κάθε τέσσερα χρόνια. Το ίδιο απέτηση ισχύει για το ΦΥΣ και για το Eurodac. Αυτό που κάναμε ήταν να φτιάξουμε ένα κοινό πλαίσιο ελέγχου που θα μπορούσε να είναι κοινό, όπως είπα, και για τις εθνικές αρχές και για την Ευρωπαϊκή Αρχή, ώστε να διενεργούν αυτό το νομικό τους καθήκον και δεν κατέστη υποχρεωτικό, αλλά θα ήταν σκόπιμο ε, τα, οι DPA να κάνουν τις επιθεωρήσεις τους σε εθνικό επίπεδο με τρόπο ώστε έτσι να μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα εφόσον τα ελέγχουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το κοινό πλαίσιο έχει δύο συνιστώσεις. Ένα, ένα, ένα πρότυπο ασφαλείας και ένα πρότυπο για τον έλεγχο των, συναγερ, των συναγερμών. Τώρα στο μέλλον θα μπορούσαμε να το, να το αναπτύξουμε περισσότερο γιατί είναι δυνατόν να, να προσθέσει κανείς πρότυπα σε αυτό το κοινό πλαίσιο. Αυτή ήταν μια δραστηριότητα λοιπόν που πήρε πολύ χρόνο, σχεδόν δύο χρόνια. Αλλά ήταν σημαντικό να στηρίξουμε τα TPA στην άσκηση των καθηκόντων τους και επίσης περιλαμβάνει μια πιο ομοιόμορφη, μάλλον οδηγεί σε μια πιο ομοιόμορφη ε, αντιμετώπιση. Επίσης οι άλλες ομάδες, το ΒΙΣ και το Eurodac εκμεταλλεύονται αυτήν την ε, δική μας δουλειά. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Άλλος ένας άξονας ο οποίος είναι μια ένα η εργασία είναι το να αυξάνουμε την ενημέρωση του κοινού. Ξέρουμε πως είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τα δικαιώματά του ώστε να μπορεί να τα ασκεί σωστά. Εάν δεν τα γνωρίζει, δεν μπορεί και να τα ασκήσει. Αυτό που σας είπα είναι ένα εργασία, δεν σταματά ποτέ. Έχουμε φτιάξει λοιπόν έναν κώδικα, έναν ε, συγγνώμη, οδηγό για τα δικαιώματα στο Σέγγεν. δίνουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ώστε να μπορεί να λάβει την, ε, την άδεια, μάλλον το αίτημα για πρόσβαση για ε, επαλήθευση ή για διαγραφή, ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες, πώς μπορούν να στραφούν στην αρχή για την προστασία των δεδομένων. Ε, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό. Ο οδηγός έχει ανέβει στα site των εθνικών αρχών αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Ε, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση δηλαδή και να επιλέξει ποιο κράτος μέλος θέλει. Αυτό είχε ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο του 2014 και έχουμε φορτώσει και μια ενημερωμένη εκδοχή του 2015. Σε αυτή την προσπάθεια την μόνιμη για την ενημέρωση του κοινού παρακολουθούμε την εκστρατεία ενημέρωση που ξεκίνησε από την Κομισιόν μαζί με τι εθνικέ αρμόδιε αρχέ σε εθνικό επίπεδο. Ελέγξαμε πώ διαδίδονται πληροφορίε και το υλικό και επίση εμεί μαζί με την DPA χρησιμοποίησαμε το site μας, τα site μας ώστε να διαδώσουμε ακόμη περισσότερο τις πληροφορίες. Κάτι ακόμα σημαντικό που κάναμε και ήθελα να το τονίσω. Ε, ε πρέπει να σας πω ότι συντηρούμε τα αρχεία του Σέγγεν. Έχουμε 20 χρόνια εργασίας. Είναι κομμάτι της ιστορίας της προστασίας των δεδομένων για την Ευρώπη. Όταν όμως το, το, Το JSA ολοκλήρωσε την εργασία του, το Συμβούλιο δεν μπορούσε πια να κάνει αυτή τη δουλειά και γι' αυτό το ανέθεσε σε εμά. Καταφέραμε να βάλουμε τα, τις πληροφορίες αυτές στη Φλωρεντία, στα Ευρωπαϊκά Αρχεία, οπότε τώρα οι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε 20 χρόνια δραστηριότητες ε, ε, των αρχών αυτών. Τώρα, για το εγγύς μέλλον. Έχουμε προτάσεις για την τροποποίηση του πλαισίου ΣΥΣ, καθώς και για την διαλειτουργικότητα. γίνει αυτό, θα, αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στα δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε συζητήσει, ήδη είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, στη, με βάση την διαλειτουργικότητα μετά από την ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά νομικώς δεν μπορούμε να, εκδώσουμε κάποια επίσημη γνωμοδότηση. Βεβαίως, Έχουμε τις απόψεις μας, αλλά έχουμε και, μία, και έναν φόβο για το... Έχουμε, έχουμε προβληματισμό όσον αφορά την αναλογικότητα, τον ε, περιορισμό των σκοπών των στόχων. Θα πρέπει δηλαδή να αιτιολογηθεί η κάθε μας επιλογή. Τώρα, τα επόμενα δύο χρόνια θα εστιάσουμε στους ε, ε, φυστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν ε, οι χρήστες για το ΣΥΣ2. Ποιος έχει πρόσβαση, για ποιο σκοπό, ποιος ελέγχει την πρόσβαση, εάν τα login αναλύονται στις χώρες, να δούμε δηλαδή τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, γιατί όπως γνωρίζετε οι χρήστες του ΣΥΣ είναι δια και διάφορες αρχές, πράγμα που σημαίνει ένα μεγάλο νούμερο ανθρώπων που έχουν πρόσβαση και είναι σημαντικό να ελέγχεται η πρόσβαση ώστε να εμποδίζεται η καταχρηστική επεξεργασία στοιχείων. Επίσης, στο πρόγραμμα εργασίας μας έχουμε την ένταξη των συναγερμών άρθρο 24. Δηλαδή πρόκειται για άρνηση προς τα άτομα να μπουν. Είναι το 90% των συναγερμών στο σύστημα. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε ποια είναι τα εθνικά κριτήρια για την ένταξη των στοιχείων εφόσον υπάρχει αυτή η νέα υποχρέωση για να λάβουμε υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Οπότε πρέπει να βάλω στο Σέγγεν για έναν άνθρωπο ε, που η βίζα του εξέπνευσε πριν από δύο μέρες, πριν μια εβδομάδα, με τον ίδιο τρόπο που θα βάλω έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, ας πούμε, είναι το ίδιο, την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να έχω απέναντι στους δύο αυτούς ανθρώπους. Πώς έγινε η αξιολόγηση αναλογικότητας. Αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε. Ε, όλα αυτά βεβαίως αφορούν την εθνική νομοθεσία και αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε θα είναι ένα από τα σημεία που θα μας απασχολήσουν και επίσης στόχο έχουμε να κάνουμε μια έρευνα όσον αφορά την αναθεώρηση των περιόδων κράτησης των στοιχείων για τις ενημερώσεις και τους συναγερμούς που μένουν για τρία χρόνια ανανεώσιμα επάπειρων μπαίνουν τα στοιχεία. Η εμπειρία μας είναι ότι οι καταχωρήσεις ανανεώνονται αυτόματα χωρίς καμία αιτιολόγηση. Ενώ τώρα ο νέο κανονισμός λέει ότι αναπερίπτωση θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και θα πρέπει να δίνεται και αιτιολόγηση για την ανανέωση ή όχι της ε, καταχώρηση. Οπότε αυτό είναι μια βασική ε, ε, αλλαγή και πρέπει να κάνουμε μια έρευνα για να διερευνήσουμε καλύτερα αυτό το τομέα. Uh, repository of best practices. This is also... Επίσης, Άλλη διαθετική εργασία είναι ότι ελέγχουμε ε, τις ε, δομές των ε, υπηρεσιών όπου πολλά κράτη-μέλη έχουμε δει ότι έχουν υποστεί περικοπές δημοσιονομικές. Και εδώ θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό αυτές οι περικοπές έχουν επηρεάσει την απόδοση του εποπτικού ρόλου των εθνικών ε, αρχών εποπτείας και κατά πόσο έχουν ακόμα τη δυνατότητα να δρουν ή αν περιορίζονται. Λόγω αυτού των περικοπών γίνονται λιγότερες επιθεωρήσεις, λιγότεροι ανθρώπινοι πόροι υπάρχουν Ίσως ε, Είναι αυτό σημαντικό και επίσης έχει να κάνει με την ανεξάρτητη φύση της εποπτείας. Γι' αυτό και θέλουμε να διερευνήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η επίπτωση των περικοπών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέρα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Επανέρχομαι σε μια ερώτηση για την δανεική υπόθεση και την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών. Σε ποιο βαθμό μάλλον εφόσον το πρόβλημα μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες μέλη. Και επειδή υπάρχει ανάθεση υπεργολαβίας εξωτερικά, δηλαδή σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις, ποιες προφυλάξεις έχετε λάβει και τι συνιστάτε εσείς. Διότι αυτό το hacking έγινε λόγω αυτής της τάσεως εμπλοκής ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. και η κυρία Ζήπελ θα είναι η πρώτη που θα λάβει το λόγο εκ των συναδέλφων μου της Εθούσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την λεπτομερή αυτή επισκόπηση του έργου σας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε και θα αντιμετωπίσετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βεβαίως και για την δήλωση στην οποία προέβητε ότι είναι σημαντικό τώρα όπου συλλέγουμε όλο και περισσότερα δεδομένα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στην προστασία δεδομένων των πολιτών. Όντω αυτό είναι σημαντικό. Έχοντα υπόψη και τις λεπτομέρειε τις οποίες αναφερθήκατε, θα προσπαθήσω να έρθω σε ορισμένες από τι πτυχέ. Μιλήσατε για την αξιολόγηση και για το γεγονό ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να αιτιολογούνται. Εάν υπάρχει ανησυχία ότι συλλέγονται υπερβολικά πολλά δεδομένα ή ότι αποθηκεύονται για μεγάλο διάστημα. Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα, δηλαδή αυτού του είδους η αιτιολόγηση, ποια μπορεί να είναι, με ποια επιχειρήματα δηλαδή αιτιολογείται την ε, μακρότερη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων. Δεύτερον, για αυτό το hacking των δεδομένων. Μιλούμε πλέον όχι για προστασία των δεδομένων, αλλά για ασφάλεια των δεδομένων. Και έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένους τομείς ε, η συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια των δεδομένων είναι σημαντική υπόθεση και ότι πρέπει να εξελίσσεται διότι Έρχονται συνεχώς νέες προκλήσεις και επομένως πρέπει να βελτιώνετε διαρκώς το σύστημά σας και υπάρχει ένα open space, υπάρχει ένας ανοιχτός χώρος. Η εντύπωσή σας είναι ότι οι διάφορες αρχές στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν συνείδηση του προβλήματος, διότι όπως είπατε, εφόσον σημειώνεται ένα πρόβλημα σε μια χώρα, τότε μπορεί τα δεδομένα όλων των πολιτών σε όλες τις χώρες να αφορούνται. Ακόμα πιο σημαντικό δε είναι η πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων. Μιλήσατε για πρόσβαση σε μια τράπεζα δεδομένων, αλλά θα πρέπει να δείτε ποιος στην ευχή έχει πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι τράπεζες δεδομένων. Πρόκληση που μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τώρα που αρχίζουμε να μιλούμε για διαλειτουργικότητα των διαφόρων τραπεζών δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εάν Εν προκειμένου σημειώνεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων που εργάζονται σε διάφορους οργανισμούς και συνεργάζονται μεταξύ των και αν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ομάδα υψηλού επίπεδου και να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα οργανωθεί στο μέλλον η διαλειτουργικότητα. Και ακόμη κάτι. Είπατε ότι είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματά του και το κοινό, διότι εφόσον δεν τα γνωρίζει δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Θεωρείτε ότι υπάρχει διάθεση εκ μέρους όλων των χωρών μελών και όλων των αρχών να συμβάλλουν σε αυτό ή σημειώνονται καθυστερήσεις διότι ναι μεν η συνειδητοποίηση από πλευράς του κοινού ίσως είναι πρόσθετο έργο και επομένως πρόσθετο βάρος και ίσως ορισμένοι να μην το κάνουν. Ποια είναι λοιπόν η εμπειρία σας σχετικά. Και άλλο ένα τελευταίο, όταν λέτε ότι επιτέλους τώρα αξιολογείτε τους συναγερμούς που σας δίνει το σύστημα. Η ερώτησή μου προκειμένου είναι πώς αξιολογείτε την αναγκαιότητα των συναγερμών για να εντάσσονται στο μέλλον, στο σύστημα και αν έχετε και άλλους εμπειρογνώμονες από άλλους χώρους, από άλλους τομείς με τους οποίους συνεργάζεστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κάρλος Κοέλιο. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ζίπελ στην έκφραση των ευχαριστειών εννοώ προς την κυρία Γκέρα και θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα της συνεργασίας των χωρών μελών. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός είναι αξιόλογος και όταν θα εγκρίνουμε το ΣΥΣ 2 γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών αρχών, γνωρίζουμε ε, ότι χρειαζόμαστε τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη για την ε, επιθεώρηση του συστήματος. Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Όμως, ταυτόχρονα, το Schengen Information System πρέπει να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του και να είναι χρήσιμο για τους σύνοριοφυλάκες και τους αστυνομικούς. Σήμερα αυτή η εποπτεία γίνεται και για το ΕΣΥΣ και για το ΒΙΣ και για το Eurodac. Ερωτήσεις. Πρώτα, ήδη η κυρία Σίπελ ανεφέρθηκε σχετικά. Θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα πρόταση για την αναθεώρηση της νομικής βάσης του ΣΥΣ, του SIS. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορική. Ερώτηση. Έχει ζητηθεί η γνώμη σα για τι διαδικασίε αυτέ. Δεύτερο. Θα υποβάλλετε έκθεση για τα εθνικά κριτήρια για την έγερση συναγερμών για πρόσωπα που έχουν αντιμετωπίσει άρνηση εισόδου. Άρθρο 24. Εγώ λέω εδώ και καιρό ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη εναρμόνιση των κριτηρίων αυτών. Όμω και για άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, για συναγερμούς, για ανθρώπους οι οποίοι ε, βρίσκονται υπό διακριτική εποπτεία. Πότε θα υποβάλλετε την έκθεση αυτή, αφού η πρόταση για την τροποποίηση του ΣΥΣ2 θα πρέπει να υποβληθεί κανονικά αρχάς του επόμενου έτους. Δεύτερο ή μάλλον τέλος, μιλήσατε για την ανάγκη να αξιολογείτε εάν οι κοινοποιήσει μετά τα τρία έτη γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των χωρών μελών έκαναν αυτόματες παρατάσεις, έδωσαν αυτόματες παρατάσεις. Δηλαδή το συναγερμό που υπάρχει μέσα στο σύστημα τον παρατείνουν αυτομάτως για τρία χρόνια. Αυτό πώς θα αξιολογείτε. Θα το κάνετε εσείς, θα το αναθέσετε εξωτερικά στις εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αξιολογήσετε όλους τους συναγερμούς, κάτι που δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν. Όλα τα αλεύτη, δηλαδή θα κάνετε μια δειγματοληπτική, ενδεχομένως επισκόπηση. Με ποια διαδικασία θα αντιμετωπίσετε το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ, Κάρλος. Δεν μου ζητεί άλλο τον λόγο. Α, η Επιτροπή, με συγχωρείτε. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ μετά την κυρία Γκέρα, να σας πω κι εγώ ότι έχουμε κάνει τα τελευταία τρία χρόνια στην δικιά μας υπηρεσία για το θέμα προστασίας δεδομένων. Τώρα ίσως και μετά η κυρία Γκέρα στο τέλος να απαντήσει σε όλα τα σχόλια. Ωραία. Ζουζάνα Γιάννησεν λέγομαι. Είμαι υπεύθυνη του τμήματος όσον αφορά το ΣΥΣ. Δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε με την κυρία Κέρα στην ομάδα συντονισμού τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και με τις χώρες μέλη, με την αστυνομία, με τις αρχές μετανάστευσης και όλες τις πτυχές του συστήματος. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεδομένων έχει τεράστια σημασία και είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται η αναλογικότητα και στο σύστημα ΣΥΣ είναι ιδιαίτερα επιτυχές και ζωτική σημασίας για τις χώρες μέλη. Η δεύτερη γενιά ΣΥΣ λοιπόν έχει ξεκινήσει υπογραμμίζοντας περισσότερο το θέμα της προστασίας των δεδομένων και αυτό μάλιστα και εξαιτία ε, της ιστορίας στη Δανία. Έλαβε χώρα πάντως με το προηγούμενο σύστημα, την πρώτη γενιά ΣΥΣ, όχι τη δεύτερη. Θα έπρεπε να κοιτάξουμε το σύστημα έτσι ώστε να το καταστήσουμε ασφαλές, να είναι προστατευμένο, λαμβάνοντα υπόψη και τις κεντρικές ε, λειτουργίες, αλλά και το τι γίνεται στις χώρες μέλη. Ο μηχανισμός αξιολόγησης έγκεν είναι πολύ σημαντικός για την προστασία του συστήματος. πηγαίνουμε στα ένσης, κοιτάμε την ασφάλεια των δεδομένων από κάθε πτυχή και την τεκμηρίωση, αλλά υπάρχει μια αξιολόγηση στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη κάθε πέντε χρόνια για το σύστημα Σέγγεν. Ένα από τα στοιχεία είναι να δούμε τι κάνουν με outsourcing οι χώρες μέλη. Κοιτάμε το ένσης, στην ανάπτυξη και τη διαδικασία outsourcing, κατά πόσο αυτή εποπτεύεται επαρκώς από τις χώρες μέλη, την κυβέρνηση, τις αρμόδιες αρχές και αν υπάρχει clearance για τα άτομα τα οποία συμμετέχουν εκεί. Συνεπώς, πολλά γίνονται από αυτού. Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή είναι η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Γιατί μόνο με καλής ποιότητας ε, δεδομένα μπορούμε να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και αυτό και με το Γιουρίκα και στις ε, χώρες μέλη και έτσι πιστεύω βελτιώνουμε την ποιότητα των δεδομένων. Αυτό το οποίο επίση κάναμε είναι ότι δώσαμε ερμηνεία από την αρχή όσον αφορά το ε, δικαίωμα πρόσβασης. Ότι υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις χώρες μέλη, ανεξάρτητα με το που υπάρχει ειδοποίηση, καταχώρηση, το alert. Μπορούν λοιπόν να υποβάλουν το αίτημά του οι αρχέ που ενδιαφέρονται και οι χώρε μέλη είναι υποχρεωμένε να απαντήσουν ακόμα και αν δεν εμπλέκεται η δικιά του χώρα. Αλλά στην διαβούλευση πρέπει να συμμετέχουν. Επίση, αναγνωρίσαμε και το θέμα της ε, ε πότε εκπνέει το σχέδιό μας. Ένα χρόνο έχουμε πει. Και πρέπει να δούμε κατά πόσο η δεκαετία ο στόχος είναι αναλογική όχι. Δεν μιλάω για άτομα, για αντικείμενα. Γιατί και τα αντικείμενα ανήκουν σε κάποιον. Άρα έχουν σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και συνδέονται με τον ε, ιδιοκτήτη βέβαια. Συνεργαζόμαστε λοιπόν συνεχώς, συμμετέχουμε σε όλες τις ομάδες σας και είμαστε ευτυχείς από τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκέρα τώρα. Να απαντήσει στους συναδέρφους παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, μετά την ιστορία στη Δανία, όπως είπατε κι εσείς, φυσικά υπάρχει πρόβλημα με το outsourcing, αλλά όχι με το outsourcing αυτό καθεαυτό, αυτό, αλλά με τον έλεγχό του. Αυτά που έγιναν στη Δανία και βρήκε ο εκεί υπόπτης δεδομένων, είναι ότι η αστυνομία δεν έλεγχε το τι έκανε ε, το outsourcing. Επίσης, ο ίδιος επεξεργαζόταν δεδομένα για το συς ε, φορολογικά, άδειες ε, ε, οδηγήσεως. Ένα σωρό δεδομένα δηλαδή πηγαίνανε σε μία μόνο εταιρεία outsourcing. Τώρα ξέρουμε τεχνικά τι ακριβώς έγινε. Πάντως, υπήρξαν μεγάλες αδυναμίες από πλευράς ασφάλειας. Με σύνδεση ίντερνετ που δεν ήταν ε, όπως έπρεπε. Όλα αυτά οδήγησαν στο να γίνει το σύστημα πιο ευάλωτο και μπορούσε να αντιγράψει ολόκληρη τη βάση δεδομένων η εταιρεία αυτή. Αυτό έγινε στο ΣΥΣ1. Τώρα έχουμε τη μεταφορά όλων αυτών στο ΣΥΣ2, που σημαίνει ότι πολλά από τα δεδομένα τα οποία έχουμε τώρα στο ΣΥΣ2, ίσως να μην είναι ασφαλή. Φυσικά υπάρχουν και πολλά νέα δεδομένα και κάποια έχουν διαγραφεί κατά την μεταφορά, αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία αντιγράφηκαν κατά τη διαδικασία αυτή στη Δανία στο ΣΥΣ 1 και που τώρα τα έχουμε και στο ΣΥΣ 2. Κανείς δεν ξέρει να πει με βεβαιότητα ποια είναι αυτά, πόσα είναι αυτά. Και τι έγινε με τα δεδομένα τα οποία αντιγράφηκαν από την εταιρεία. Πουλήθηκαν όλα, κάποια. Υπάρχουν τρίτα μέρη που έχουν μέρος των δεδομένων αυτών. Ίσως να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν αρκετές για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι έχει γίνει με όλα αυτά τα δεδομένα. Πάντως για τα outsourcing θέλω επίσης να τονίσω ότι τώρα υπάρχει αξιολόγηση του Σέγγεν, γίνεται αυτή την εποχή και υπάρχει μια ερώτηση στην αξιολόγηση αυτή για το outsourcing και για το πώς ελέγχουν τους outsourcers αυτούς οι χώρες μέλη. Τι προνόμια έχουν σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων. Για να δούμε κατά πόσο οι χώρες ε, μέλη ελέγχουν ή όχι το τι κάνουν με τα δεδομένα αυτά οι εταιρείε που έχουν αναλάβει ως outsourcing. Αυτή τη φορά με το πρόβλημα που είχαμε δεν έφταιγε ένα συγκεκριμένο έφταιγε το γεγονός ότι δεν υπήρχε έλεγχος. Επειδή λοιπόν είναι επόπτες δεδομένων οι χώρες μέλη, έχουν την ευθύνη να ελέγχουν και να ξέρουν ανα πάσα στιγμή τι έχει γίνει με τα δεδομένα. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια τόσο ευαίσθητη βάση δεδομένων, οι χώρες μέλη θα έπρεπε να προσέχουν πάρα πολύ σε ποιες εταιρείε δίνουν outsourcing. Και εννοείται ότι πρέπει να ελέγχουν. Δεν μπορεί τον έλεγχο να το κάνουν οι εταιρείε outsourcing. Για την κυρία Σίπελ. λέτε ότι δεν υπάρχει επαρκή συνειδητοποίηση για τα θέματα ασφάλειας. Αυτό ισχύει τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς βέβαια οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά για την ασφάλεια τράπεζες για παράδειγμα για την ασφάλεια δεδομένων και κάποιες δημόσιες αρχές ε, τελικά μερικές φορές πρέπει να γίνει κάποια παραβίαση για να ξυπνήσει ο κόσμος και να αποφασίσει να επενδύσει σε προσωπικό, σε ειδικού συνεργάτες. Οπότε σίγουρα χρειάζεται περισσότερη συνειδητοποίηση. Και η δικιά μας η δουλειά και το δικό μας το καθήκον είναι να τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια για τα δεδομένα. Είτε πρόκειται για τα προσωπικά δεδομένα, είτε για τη συνειδητοποίηση πάντα. Θα υπάρχει μια ιστοσελίδα για το κοινό. Ρωτήσατε αν οι δημόσιες αρχές βρίσκονται όλε στην ίδια σελίδα. Γιατί πολλές φορές λέμε δεν πρέπει να δημοσιεύσουμε πολλά, γιατί τότε θα πλημμυριστούμε από σχόλια. Εμείς επενδύουμε το χρόνο μας στα θέματα Σέγγεν εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε πληροφορίες και σε πολλές γλώσσες. Ανάλογα με το ποιοι υπήκοοι τρίτη χώρας μας προσεγγίζουν περισσότερο. Έχει γίνει λοιπόν αρκετή δουλειά από αυτού. Και επίσης η ομάδα θα βοηθήσει πολύ εδώ, γιατί θα έχει και τη δικιά της ιστοσελίδα. Όλα τα θέματα δραστηριοτήτων μας θα αναρτηθούν λοιπόν και εκεί. Ρωτήσατε επίσης για την ανανέωση των ε, καταχωρήσεων, των alerts, ο κύριος Σκόγιο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να το ψάξουμε. Τα στατιστικά δεδομένα βοηθούν λιγάκι για να προχωρήσει κανείς. Θα αρχίσουμε λοιπόν με στατιστικά δεδομένα, να δούμε πόσες τέτοιες καταχωρήσεις ανανεώνονται, πόσο συχνά και μετά όπως γίνεται σε κάθε επιθεώρηση θα ελέγχουμε κάθε τόσο Φυσικά όχι και τις χιλιάδες καταχωρήσεις, αλλά ένα μέρος έτσι ενδεικτικά. Και θα ζητάμε την αιτιολόγηση, γιατί τώρα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Βέβαια Όλα έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα που είναι πολύ βασική αρχή. Οι καταχωρήσεις αυτές, τα LEDS, πρέπει να καταχωρούνται και να κρατιόνται όσο είναι αναγκαίες. Δεν χρειάζεται να μένουν τρία χρόνια, αλλά την αξιολόγηση δεν την κάνει ο επόπτης ε, δεδομένων ο Ευρωπαίος, αλλά οι εθνικές αρχές. Η αξιολόγηση πάντως που γίνεται πρέπει να αιτιολογείται. Για μας είναι σημαντικό να ελέγχουμε κατά πόσο υπάρχει αιτιολόγηση. Γιατί το συγκεκριμένο άτομο πρέπει να παραμείνει στο σύστημα. Αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση από τις χώρες μέλη, τότε θεωρούμε ότι τελείωσε. Δεν χρειάζεται να είναι στο σύστημα το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν εφ' εξής. Όσον αφορά τώρα τα εθνικά κριτήρια, κύριε Κόγιο Φοβάμαι ότι αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά για να συνεισφέρουμε στις προτάσεις. Τα πρώτα χρόνια δραστηριοτήτων το κάναμε για να βοηθήσουμε για μια έκθεση που έπρεπε να ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τρία χρόνια. Αλλά πήρε πολύ χρόνο. Και έτσι δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να πας όλες τις χώρες μέλη και να τα ψάξεις. Υπάρχει το άρθρο 24 που λέει για ποιους λόγους μπορείς να δημιουργήσεις μια καταχώρηση, να βάλεις κάποιον στο σύστημα, δηλαδή αν υπάρχει έγκλημα, αν υπάρχει κίνδυνος για έγκλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια καταχώρηση στο σύστημα και πρέπει να περνάμε από την εθνική νομοθεσία κάθε φορά και να βλέπουμε τι είναι κοινό μεταξύ μας και τι όχι. Και όταν έχουμε κάνει αυτή την επιθεώρηση, μετά μπορούμε να δούμε προς τα που πρέπει να πάμε. Και η πρότασή σας να έχουμε περισσότερο εναρμονισμένα κριτήρια φυσικά και θα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήταν τέλειο, γιατί έτσι θα μπορούσαμε πιο εύκολα να κάνουμε τους ελέγχους και να αποφεύγουμε το θέμα της αναλογικότητας ε, με τις καταχωρήσεις. Και όπως έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα της ποιότητας, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μερικές φορές έχετε σε μία καταχώρηση ένα-δύο ονόματα. Αν είναι από κάποιο σημείο του κόσμου που έχει εκατομμύρια ανθρώπους, έχετε το ίδιο όνομα πάρα πολλέ φορές. Αν έχετε μόνο τα ονόματα και δεν έχετε τίποτα άλλο, καμιά φορά έχετε και ημερομηνία γέννηση καμιά φορά το κάνει αυτό. Αν λοιπόν έχετε μόνο όνομα, δεν μπορείτε να αποφασίσετε για ποιον ακριβώ πρόκειται. Στα σύνορα ε, σταματάτε ανθρώπους με αυτό το όνομα, παρόλο που δεν είναι αυτοί που πρέπει να σταματήσετε. Οπότε και δημιουργείται άλλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Στην Πορτογαλία, από όπου προέρχομαι κι εγώ, έχουν υπάρξει πάρα πολλά αιτήματα, όλοι πάνε στον επόπτη και αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα καθημερινά. Δηλαδή ότι σταματάμε ανθρώπους που δεν είναι αυτοί που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα λόγω συνωνυμίας. Οπότε θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα έχουμε καταφέρει έγκαιρα. Έρχομαι σε μια άλλη ερώτησή σας για την ε, πρόκληση της διαλειτουργικότητας και αν ε, συμμετέχουμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου ή απλώς γνωμοδοτούμε. Όπως ε, είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε καλή θεσμική σχέση με την Επιτροπή. Καλούμε την Επιτροπή να έρχεται στις συναντήσεις μας κάποια συγκεκριμένη στιγμή για να μας ενημερώνει. Ρωτάμε πράγματα και η Επιτροπή μας εξηγεί. Οπότε αυτή η σχέση είναι καλή. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη συμμετοχή. Είναι θετικό, αλλά επίσημα δεν μας ζητούν γνωμοδότηση. Δηλαδή μπορεί στην πράξη να ανακατευόμαστε, αλλά όχι επίσημα. Ενώ όλα τα θέματα ΣΥΣ ε, θα έπρεπε να εμπλέκουν όλες τις εθνικές εποπτικές αρχές. Είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε γιατί τα προβλήματα που έχουμε με το τρέχον σύστημα και με τα άλλα ξέρουμε ήδη σε εθνικό επίπεδο πότε είναι ολοκληρωμένα ή όχι αυτά τα συστήματα για μία ε, ενιαία αντιμετώπιση της ε, προκειμένου να βρούμε μια αρχή συμμόρφωσης και τι δικαιώματα έχουν. Μερικές φορές σε κάποιες χώρες ισχύει, αλλά σε άλλες όχι. Με αυτό που λέμε single search, δηλαδή ψάχνω ένα όνομα, αν ε, έχω προνομιακή πρόσβαση, μπαίνω στο σύστημα. Τα συστήματα δεν είναι διαλειτουργικά, είναι χωρισμένα το ένα από το άλλο, αλλά μπορώ με αυτό το single search να ψάξω σε όλα τα συστήματα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από πλευράς ε, αυτού που πρέπει να ψάξει, είναι τεράστιο κέρδος χρόνου. Συμμετέχουμε λοιπόν στις συζητήσεις, αλλά επίσημα, όπως σας είπα, δεν έχουμε αυτό το καθεστώς. Θέλουμε όμως. Αν εξαρτάται από εσά, σας λέω ότι θα το θέλαμε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέρα για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να συνοψίσω αυτό το θέμα. Την επόμενη Δευτέρα ο κύριος Ζούτα θα πάει στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου. Έχουμε την νέα ομάδα εργασίας της ΛΥΜΠΕ όπου οι συντονιστές ε, θα επικεντρώσουν πολύ την προσοχή τους. Ο κύριος Κοέγιο προεδρεύει αυτή την ομάδα εργασίας ώστε να συνεχίζεται ο έλεγχος του Σέγγεν. Επίσης έχουμε και την αποστολή της Επιτροπής μας 3 και 4 Νοεμβρίου στο Εουλίσα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γέρα για την παρουσία σας λοιπόν εδώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Uh, λοιπόν, προχωράμε τώρα στο σημείο 20, κύριε Δεπρέ, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχουμε το ίδιο θέμα. Έχετε καταθέσει μια ε, ερώτηση στην Επιτροπή και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει γέρος απαντήσει η Επιτροπή υπό τον, υπό τον κανόνα 30 του κανονισμού καλούμε την Επιτροπή εδώ και τίθεται το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εσείς λοιπόν καταθέσατε αυτή την ερώτηση ε, για τις αποφάσεις επιστροφής και τα μέτρα απομάκρυνσης, αν καταγράφονται στο ΣΥΣΙ στο Eurodac. Έχετε θέσει την ερώτηση λοιπόν από τις 15 Σεπτεμβρίου και λήψη απάντηση ζητήσατε να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Ντεπίρα θα σας δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Τζεράρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν πειράζει που αργήσαμε γιατί η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα. Ε, είχα θέσει λοιπόν πριν λίγο καιρό μια ερώτηση στην Επιτροπή ρωτώντα αν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια βάση δεδομένων ή ένα διάβλο ανταλλαγή πληροφοριών που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να γνωρίζουν κατά πόσο ένα λοδαπό ε, Ε, χωρίς ε, ε, άδεια παραμονής μπορεί να είναι καταγεγραμμένος κάπου, σε κάποια βάση δεδομένων. Η Κομισιόν είπε πως δεν έχει τέτοια βάση δεδομένων, αλλά είπε ότι θα προτείνει να καταστεί υποχρεωτική εγγραφή στο ΣΥΣ. Μπορεί να μας διευκρινίσει η Κομισιόν, να μας πει γιατί το ΣΥΣ είναι το καλύτερο μέσο να καταγραφούν αυτού του είδους τα μέτρα Απομάκρυνση ή επιστροφή, γιατί παράλληλα η Κομισιόν έχει καταθέσει πρόταση που στόχο έχει να καταστήσει υποχρεωτική την εγγραφή στο Eurodac από πλευρά των 100 μελών όλων των ε, ε, παράνομων ε, λοδαπών, δηλαδή που δεν έχουν χαρτιά, σε μια βάση δεδομένων που αρκετά μεγάλη. Αλλά σε τι θα χρησιμεύσει εφόσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή τους αφού δεν έχουν έχουν λάβει ε, ε, εντολή να φύγουν ε, ή να καταλήψουν την επικράτη, πώς Τι, τι ενδιαφέρον έχει να γράφονται όλα αυτά στο Γιουροντακ, αφού δεν θα έχουμε πληροφορίες για αυτούς τους ανθρώπους. Βέλκερ Γιάνσεν είναι εδώ για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Ντεπρέ. Καταρχά, θα ήθελα να σα διαβάσω την απάντηση στην πρώτη ερώτηση, που ήταν η 48. 44-2016 που και κρίθηκε επισήμω από την Κομισιόν και λέει τα εξή. Οι κανόνε και οι διαδικασίε σε σχέση με την απομάκρυνση τρι, ε, πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν ε, αντικανονικά στην Ένωση διέπονται από αυτήν την οδηγία. Η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσο ο κανόνα αυτό ε, απαντά στι προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ω αποτέλεσμα τη ε, εισρωή μεγάλου αριθμού μεταναστών καθώς και στην Ευρώπη και τη δευτερεύουσα του μετακίνηση εντός Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν συλλέγουμε τέτοια στοιχεία. Είναι λοιπόν δυνατόν ένα αντικανονικό ε, μετανάστη που έχει νομική υποχρέωση να φύγει, να αποφύγει την επιστροφή απλώ μετακινούμενο προς άλλο κράτο μέλος εντός της ζώνης ε, Σέγγεν. Εάν συλληφθεί θα πρέπει να ξεκινήσει νέα διαδικασία για την επιστροφή του εν λόγω ανθρώπου. Ε, για η Κομισιόν ε, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταγράφει τις πληροφορίες αυτές στο ΣΥΣ ε, ε, και να καταστήσει υποχρεωτικό για τα κρατημέλη να καταγράφονται όλες οι είσοδοι στην επικράτειά τους και έτσι θα δίνονται ειδοποίηση μέσω του Σέγγεν για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τους παρανόμους αυτούς μετανάστες. Πράγμα που θα ενισχύσει τις πληροφορίες που έχουμε για τους ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν μετακινούμενοι σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα χρειαστεί νομικές και τεχνικές αλλαγές στο ΣΥΣ, αλλά θα αυξήσει και την εναρμόνιση και τη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές που, για την, αρμόδιες για την επιστροφή. Και αυτό είναι απάντηση για την πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση που έφτασε στις 31 Αυγούστου. Ζητώ συγγνώμη ε, ε, που καθυστερήσαμε με την επίθυνση μια μας από απάντηση. 17 Οκτωβρίου υιοθετήθηκε. 7 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Το ΣΥΣ επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο μέτρο, μάλλον εργαλείο, όπου να καταγράφονται οι αποφάσεις επιστροφής. Το ΣΥΣ είναι ο ο η ευρύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη και είναι άμεσα διαθέσιμη στην πρώτη γραμμή των αστυνομικών ερευνών και των συνοριοφυλάκων όπου μπορούν άμεσα να προβούν στις ενέργεια που απαιτείται. Δεν ε, ισχύει αυτό για το Eurodac που έχει πολύ περιορισμένο σκοπό και στηρίζει βασικά την εφαρμογή κανονισμού του Δουβλίνου. Επίσης, ε, το πεδίο του Eurodac δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για επιστροφές. Ας πούμε, δεν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις για επιστροφές που έχουν να κάνουν με εγκληματίες και γι' αυτό είναι καλύτερα να περιλαμβάνονται στο ΣΥΣ. Εκεί περιλαμβάνονται ήδη τα όσα αποφασίζονται από το άρθρο 24 του κανονισμού για το ΣΥΣ. Τα όσα θα προσθεθούν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη μετά από την προηγούμενη φάση, όπου οι επαγορεύσεις εισόδου ήδη ε, γίνονται μέσω μιας προηγούμενης γραπτής απόφασης. Άλλη σημαντική εξέλιξη για το ΣΥΣ. Μου ζήτησαν οι διερμηνείς να μιλήσετε λίγο πιο αργά όταν διαβάζετε τις αποφάσεις σας λέει ο Δεπρέ. Βασικά πιστεύω πως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για το ΣΥΣ, γιατί είναι ε, το πιο ευρύ ε, μέσο ανταλλαγής πληροφορίων, ήδη το έχουν στη διαθεσή τους δηλαδή αστυνομικοί, που μπορούν να προβούν στις ενέργειες που χρειάζεται άμεσα, πράγμα που δεν συμβαίνει με το Eurodac, γιατί το Eurodac έχει πολύ συγκεκριμένο περιορισμένο σκοπό, αποθηκεύει τα στοιχεία των ετούντων άσυλων καθώς και των ε, παράνομων μεταναστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικές περιστάσεις από εγκεκριμένους χρήστες, αλλά όχι στην κλίμακα του χρήσης του ΣΥΣ. Όταν ελέγχεται ένας άνθρωπος λοιπόν, Οι αστυνομικοί μέσω των ειδοποιήσεων του ΣΥΣ μπορούν να προβούν σε ενέργειες. Αυτό είναι το πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το πεδίο του Eurodac δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που μπορεί να είναι αντικείμενο απόφασης επιστροφής επειδή δεν περιλαμβάνεται η γραπτή ε, ποινή ε, στο Eurodac. Ενώ περιλαμβάνεται στο ΣΥΣ μέσω υπό τη μορφή τη απαγόρευση εισόδου και ξέρετε ότι το σύστημα ΣΥΣ καλύπτει ήδη τι απαγορεύσει εισόδου. Είναι το στάδιο όπου κανείς φεύγει από την επικράτεια Σέγγεν, τότε εκδίδεται απαγόρευση εισόδου. Ε, Φόσον λοιπόν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει, θα πρέπει να είναι αντικείμενο επιστροφής και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστραφεί ε, αυτός ο άνθρωπος. Ε, το ΣΥΣ για την ώρα δεν το βλέπει αυτό το στάδιο της επιστροφής, βλέπει μόνο την φάση όπου ο άνθρωπος φεύγει αλλά δεν πρέπει να ξαναέρθει, δεν πρέπει να, να το επιτρέπει να επιστρέψει φυσική λοιπόν εξέλιξη ώστε να συμπεριληφθεί και μια προηγούμενη φάση της ε, διαδικασίας επιστροφής. Αυτό που επίσης είναι σημαντική εξέλιξη στο ΣΥΣ είναι ότι προστίθεται μια λειτουργικότητα αυτόματης αναγνώρισης τελικών αποτυπωμάτων που θα προσθεθεί ε, συντόμως, ώστε οι άνθρωποι που έχουν πολλαπλές ταυτότητες ή, ή πλαστές ταυτότητες να αναγνωρίζονται επί τη βάση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων τους. Φυσικά, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν υπό ποιες συνθήκες ε, ε, μπορεί να γίνει έλεγχος για την επιστροφή. Πάντως είναι βασικό στοιχείο του ΣΥΣ να εντοπίζει τους παράνομους μετανάστες. Ακόμη και εγώ κάπω τάχασα σε όλα αυτέ τι εξηγήσει. Θέλει, Ζεράρ, να ζητήσει ευκαιρία. Παρακαλώ, είναι δική σου ερώτηση. Α, λοιπόν, αν στο ΣΥΣ έχετε και θα έχετε ένα σύστημα αναγνωρίση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, γιατί να επιβληθεί σε όλα τα κρατημέλη να συλλέγουν όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα όλων των παράνομων μεταναστών που έχουν στην επικράτειά του. Σε τι θα χρησιμεύσει αυτό. Προσπαθούμε, λέει ο Πρόεδρος, και να ικανοποιήσουμε τον κύριο Ντεπρέ και θα μείνουμε εδώ μέχρι που να το απαντήσετε. Αλλά λίγο αργά να μιλάτε πάντως ε, απαντώντας. Ναι, μάλιστα. Για την ώρα μπορεί κανείς μόνο να αναζητήσει στο ΣΥΣ έναν άνθρωπο από το, με το όνομα και την ε, ημερομηνία γέννησής του. Αν ένας άνθρωπος χρησιμοποιήσει πλαστή ταυτότητα, ακόμα και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ενταγμένος στο σύστημα, δεν θα βρεθεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα αναζήτησης ε, μέσω δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αν λοιπόν οι μετανάστες ε, φεύγουν από τη χώρα όπου έκαναν έτοιμα ασύλου και πάνε σε άλλη χώρα για να ζητήσουν και εκεί άσυλο, ή, αλλά με άλλα χαρτιά και άλλη ταυτότητα, στο ΣΥΣ είναι δυνατόν να εντοπιστούν επί τη βάση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων και καθώ επίση θα φαίνεται αν είναι αντικείμενο απόφασης επιστροφή. Εγώ επανέρχομαι στην ερώτησή μου. Γιατί θα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να, ζητάνε ανθρωπιστικά αποτυπώματα και ε, αναγνώριση ε, προσώπου όλων των μεταναστών, εφόσον θα μπορούμε να το κάνουμε αύριο μεθαύριο από το ΣΥΣ. Ε, that basically fundamentally Eurodac and the SIS they have a να σας πω ότι το ΣΥΣ και το Eurodac έχουν διαφορετικό σκοπό. I, uh, asylum seeker and irregular migrant and also... Το ΣΥΣ ε, θέλει να εντοπίζει τους παράνομους μετανάστες αλλά και να βλέπει πού έχουν καταγραφεί πρώτα και ποια χώρα είναι υπεύθυνη για να κάνει την διαδικασία ασύλου. Στο, στο Eurodac, με συγχωρείτε. Είναι πολύ περιορισμένο δηλαδή η χρήση και εκεί αποθηκεύει το Eurodac μόνο τα θεχθλικά αποτυπώματα για την ώρα. Όμως το ΣΥΣ έχει άλλο στόχο. Με το ΣΥΣ οι αστυνομικοί επιτόπου μπορούν να προβούν σε άμεσες ενέργειες. Όχι μόνο να εντοπίσουν και να βρουν έναν άνθρωπο και να τον ελέγξουν, αλλά να προβούν και σε δράση. Είτε να τον συλλήψουν, συλλάβουν, είτε να τον προστατεύσουν, αναλόγως τι γίνεται εν λόγω στην περίπτωση. Η χρήση του ΣΥΣ λοιπόν είναι διαθέσιμη για κάθε αστυνομικό. Στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη γραμμή των συνοριακών ελέγχων. Όταν υπάρχει ανάγκη για εντοπισμό ενός ανθρώπου υπάρχει το ΣΥΣ. Γι' αυτό το ΣΥΣ είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να αποθηκευθούν οι πληροφορίε για τι αποφάσει επιστροφή. γιατί επί τόπου οι αστυνομικοί όταν ε, ανακρίνουν έναν άνθρωπο θα μπορούν να, να ε, βρουν την ταυτότητά του άμεσα και να την επαληθεύσουν. Τελείω διαφορετική σκοπή των δύο συστημάτων. Εγώ κατάλαβα τι λέει. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο. θα επανέλθω δερμύτερος. Okay, um, Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνουμε το νόημα της απαντήσεώς σας. Μιλάτε για τις διαφορές των δύο τραπεζών δεδομένων. Ο Ντεπρέ ρωτά γιατί δεν τα βάζετε στο Eurodac. Δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση. Θα θέλετε λοιπόν να ε, συνεχίσετε να το ψάχνετε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς παρακαλώ ε, πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα. Το Eurodac δεν είναι πλήρης τράπεζα δεδομένων για τη μετανάστευση. Είναι ένα σύστημα αρχείου. Δεν βάζει το ιστορικό μέσα. Μόνο τα δακτυλοσκοπικά αποτυπώματα του μετανάστη. Ούτε και στο άλλο σύστημα υπάρχει ιστορικό, αλλά υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στο SIS. Και πιο σημαντικό ακόμη υπάρχει μια συγκεκριμένη δράση που δεν διαθέτει το Eurodac. Και υπάρχει ολόκληρη υποδομή πίσω από το SIS με συμπληρωματικές πληροφορίες. Ενώ Εκεί μπορεί μάλιστα να βρεθεί ολόκληρο το ιστορικό των κινήσεων του συγκεκριμένου προσώπου για να μπορούν οι αρχές να λάβουν την κατάλληλη δράση. Αυτό δεν συμβαίνει με το Eurodac, διότι το Eurodac έχει πολύ περιορισμένο σκοπό χρήσεως και βεβαίω πολύ διαφορετικό σκοπό γενικώ. Θα το αφήσουμε για την ώρα το θέμα αυτό, λέει ο πρόεδρος ε, Μωράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ή μάλλον έχω να πω το εξής. θα επανεξετάσουμε το ΣΥΣ 2, και Eurodac και θα διαθέσουμε αρκετό χρόνο στα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας. Άρα πολύ σύντομα θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ Γεράρ, και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέμα 22. αποστολή της Επιτροπής Λίμπε στην ΕΑΣΟ στην Μάλτα στα μέσα Ιουλίου του 2016 εξέταση σχεδίου έκθεση της αντιπροσωπείας. 18 έως 20 Ιουλίου λοιπόν οι συνάδελφοί μας της Λίμπε πήγαν στην ΕΑΣΟ, στο γραφείο της ΕΑΣΟ δηλαδή, η Σεσίλ Κιένγκε ήταν ε, μαζί τους, καθώς και άλλοι συναδελφοί μας, ο αυτόν ο κ. στα πλαίσια της αναδιετία ε, επισκέψεως της Επιτροπής μας στον ΕΑΣΟ, βεβαίως για την εξέταση θεμάτων μετανάστευση και προσφύγων. Λοιπόν, έχουν το σχέδιο εκθέσεως. Σεσίλια, ε, έχετε εσείς τον λόγο, ορίστε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, ε, μας υποδέχθηκαν πολύ θερμά και με μεγάλο επαγγελματισμό. Μας υποδέχθηκε ο Ιωσέ Καρέρα, ο διευθυντής του ΙΣΕΑΖΟ καθώς και οι Μαλτέζικε Αρχές, γιατί μπορέσαμε να συναντήσουμε και τις αρχές της Μάλτας, καθώς και εκπροσώπους της Κοινωνία των πολιτών. Από τις επαφές που είχαμε με όλους τους εκπροσώπους του ΣΕΑΖΟ ε, προέκυψε μεγάλος επαγγελματισμός με τον οποίο ε, ασκούν τα καθήκοντά τους. Ε, καθήκοντα τα οποία ξεπερνούν τον θεσμικό αναγνωρισμένο τους ρόλο, να θυμίσω ότι η ΑΖΟ συνέβαλε στην, ε, στο άνοιγμα γραφείων ε, της πρώτης γραμμής στη Βουλγαρία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Δεν ε, υπάρχει όμως αρκετό προσωπικό. Είναι μικρό το γραφείο, ότι το αποσπασμένο, αποσπασμένο προσωπικό είναι από τα κράτη-μέλη και είναι λειτουργικό σε πολύ μικρό βαθμό. Για να μην πω για το προϋπολογισμό που είναι τελείως τελείως ε, ανεπαρκές. Η εργασία της, ε, αυτή έχει γίνει στην Ελλάδα με ε, εξαιρετική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Τον, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο έφτασαν στην Ελλάδα χιλιάδες άνθρωποι από τη Συρία και στο πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία οι αρμοδιότητε του ε, περιορίζονται στο να δίνουν πληροφορίες στις ελληνικές αρχές για το κατά πόσο είναι αποδεκτέ οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Ε, η ΑΖΟ έχει επίσης υποστηρίξει στην ε, τις συνεντεύξεις που γίνονται στους ετούντες άσυλο, που είναι διαφορετικοί από εκείνους που έχουν άλλο καθεστώς, όπως οι πολίτες του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν. Μετά από αίτημα των αρνητικών αρχών, η ΑΖΟ ανέλαβε την προκαταχώρηση που είναι το πρώτο βήμα προς την διαδικασία ασύλου, καθώς και να στηρίξει το πρόγραμμα της επανεγκατάστασης. Ο Διευθυντής Ιωσέ Καρέρα είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στήσε μία υψηλού επίπεδου ε, αποστολή για να τονιστεί συνεργασία ανάμεσα στα κατημέρια και να στηριχτεί, γιατί πολλές φορές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές και πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα θέματα της ασφάλειας. Ο ρόλος της ΕΑΖΟ ήταν σημαντικός και στην Ιταλία. Το πρώτο τμήμα ήταν αυτό που αφορούσε την Ιταλία, το δεύτερο όμως αφορούσε την Ιταλία για τη φάση της καταγραφής των μεταναστών. Επίσης είναι σημαντικός ο ρόλος της στις τρίτες χώρες, για παράδειγμα στα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Όσον αφορά τώρα την επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση προς από την Τουρκία, υπήρξαν περισσότερες μετεγκαταστάσεις από ό,τι επαναπατρισμοί. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον υπεύθυνο του Τμήματος Ανάλυση και Ενημέρωση. Μας είπαν ότι η ΑΖΟ δεν δίνει εξολογήσεις για την ασφάλεια των χωρών προέλευσης ή των ασφαλών χωρών, αλλά συλλέγει μόνο ουδέτερες πληροφορίες και Αντικειμένικέ πληροφορίε για τι διάφορε χώρε. Η έκθεση για την ενημέρωση για τι χώρε προέλευση συνδέεται με το προσωπικό τη ΕΑΖΟ και σε συνεργασία με εμπειρογνώμες από τα κάτι Ο νέο κανονισμό, ωστόσο, θα επεκτείνει τις αρμοδιότητες ΕΑΖΟ για την ανάλυση στην κατάσταση τη χώρα προέλευση. στη στιγμή που τα κατημέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την ανάλυση στην εφαρμογή των μέτρων διεθνού Προστασία. Έπειτα, κάποια ειδικά θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ήταν το θέμα της κατάρτισης και είχαμε και μαρτυρίες για το ρόλο που έχει παίξει η ΆΖΟ στην κατάρτιση των καταρτιστών διαπιστώσαμε, τη ε, μάλλον συζητήσαμε το δραματικό θέμα των ανηλίκων και του εμπορίου ανθρώπων και τον επαγγελματισμό με τον οποίο το προσωπικό της ΕΑΖΟ προσφέρει ε, κατάρτιση στα προσωπικό στο, στο των μελών. Επίσης το ΕΑΖΟ θα ασχοληθεί με τα θύματα των βασανιστήριων. Επίσης με τον Διευθυντή μιλήσαμε για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει η ΕΑΖΟ όταν θα γίνει ε, οργανισμός αυτό καθ' αυτό. Επίση, ο Διευθυντή τόνισε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πρόσβαση σε διάφορε ε, βάσει δεδομένων που θα επιτρέψει τη χρήση των μεταδεδομένων για να ορίζονται καλύτερα και αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ισχύουσε καταστάσει. Ε, για την ΕΑΖΟ θα πρέπει να δούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε η υπηρεσία αυτή να έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό και ε, προπολογισμό, συγγνώμη, και το κατάλληλο προσωπικό. Συζητήσαμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών της Μάλτας και σταθήκαμε στην ανάγκη βελτίωσης του μηχανισμού μετεγκατάστασης, καθώς ε, και την ανάγκη ε, χάραξης με, ε, κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Ήταν πολύ ανθρώπινη αλλά και πολύ επαγγελματική η δική μας αποστολή. θα σε επαφή με ανθρώπους που κάνουν δύσκολη δουλειά ε, και που θέλουν ε, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ε, ανεξάρτητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητή κυρία Κιένγκε για την εκθεσή σας. Την εκτιμούμε ιδιαίτερως. Άλλοι δύο συνάδελφοι πήγαν μαζί και θα ήθελα να λάβουν το λόγο. και Ο Σκουέλιο είναι ένας από αυτούς. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Κιένγκε. Πήγα μαζί με τις κυρίες Κιένγκε και Στέβενς και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δύο-τρία σχόλια. Πρώτα συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Κιένγκε. Πρώτον, η ΕΑΣΟ και ο διευθυντής της Κάνουν πραγματικά θαυμάσια δουλειά. Δεύτερο, η ΆΣΟ στερείται προσωπικού και χρηματοδοτήσεων και οι αρμοδιότητες της δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσει τα όσα απαιτούνται. Τρίτο, προσωπική μου γνώμη αυτή, είναι σαφές για μένα ότι οι χώρες μέλη χρειάζονται την ΕΑΣΟ, αλλά δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να την εξοπλίσουν με τα αναγκαία. Αυτά τα σχόλια μου επιτρέπουν να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί σωστά η νέα νομική βάση και να βελτιωθεί το δυνατόν συντομότερα η κατάσταση της, του νέου οργανισμού ασύλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, πολύ ξεκάθαρα πράγματα και σε πολύ σύντομο χρόνο τα είπατε. Είμαι βέβαιος ότι η ΕΑΣΟ θα συμφωνήσει. Και ο κ. Χάλα Άχο θα μιλήσει ως κυρία Χέργια Στίβενς. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Θα διαβάσω με την άδειά σας το μήνυμα της κυρίας Στίβενς. Λέει λοιπόν η κυρία Στίβενς, είχα το μέγα προνόμιο να με σκεφτώ την ΕΑΣΟ μαζί με τους αδέρφους μου και είδα πόσο δρώνουν κάτω από μεγάλη πίεση. Είναι σαφές ότι έχει έρθει η ώρα τους, διότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια πίεση. Εγώ γενικώ δεν είμαι υπέρ της διευρύνσεως των ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά για, στην περίπτωση της ΕΑΣΟ είναι σωστό. Χρειάζεται δηλαδή περισσότερη χρηματοδότηση για επάνδρωση καθώς και για ε, εκπαίδευση. Είναι απαιτητικό το έργο της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές και να μπορέσει να διακρίνει τους πραγματικούς πρόσφυγες, αυτούς που πετούν άσυλο και αυτούς που απλώς επιθυμούν να διέλθουν τα σύνορα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη ενίσχυση ο οργανισμός αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς. Εφόσον όχι, ευχαριστώ την κυρία Κι Ένγκε για τα όσα εξήγησε για την σημαντική αυτή επίσκεψη καθώς και την έκθεσή της που βεβαίω θα λάβουμε ως βάση για το έργο μας για την ΕΑΣΟ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι και βεβαίως σημειώνουμε τα όσα μας εξηγήσατε. Τώρα θα θέλαμε να προχωρήσουμε κυρίε και κύριοι στο 21. Πάλι θέμα ασύλου. Πρόκειται για γνωμοδότηση για την αντιμετώπιση μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών και για τον ρόλο της εξωτερικής δράσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρόκειται για την γνωμοδότηση της κυρίας Βεργία Κριστίν. Σύντομη εισαγωγή πριν λάβει το λόγο η Μαρή Κριστίν για να κάνει την εισαγωγή στην έκθεσή της. Στις 7 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση η ανακοίνωση αυτή υπευλήθη στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο του 2016 και αναλάβαμε να κάνουμε γνωμοδότηση για λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών. Οι συντονιστές της 11 Εβδόμου αποφάσισαν να αναθέσουν την ε, γνωμοδότηση στην πολιτική ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς και την εισήγηση ανέλαβε η κυρία Βερζιά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα προσθέσω κάτι και εγώ στην εισαγωγή αυτή. Μεταξύ άλλων, έχω αναλάβει στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μια έκθεση που την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να υιοθετηθεί για τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Φυσικά και έχω διαβάσει με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση ΑΦΕΤ ΔΕΒΕ των συναδάλφων Βαλενθιάνο και Ντίαθ Ντεμέρα και σε πολλά συμπίπτει η έκθεση που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα με την έκθεση αυτή ΔΕΒΕ ΑΦΕΤ. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση από αυτού. Το να κάνει κανείς ε, μια γνωμοδότηση με 1500 γράμματα, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Ε, με τους σκιώδεις ηγητές το συζητήσαμε, τους εξήγησα την κατάσταση. Το σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν που σας υποβάλλω, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάπως κουτσό. Σίγουρα χρειάζονται και διάφορες αποχρώσεις αυτό, αλλά νομίζω ότι τα κύρια ζητήματα τα έχω συμπεριλάβει προσπαθώντας να επικεντρωθώ στα θέματα αρμοδιότητας της ε, ΛΥΜΠΕ και στις ανησυχίες που έχουμε εμείς ε, εν ώψη των ευρωπαϊκών πολιτικών επί του θέματος. Καταρχήν, κάνω διαπίστωση. με 500.000 εκριζωμένους ανθρώπους. Η ύπατη αρμοστία χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο και για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες λίγο πολύ. Εκφράζω την αλληλεγγύη που πρέπει να επιδεικνύουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να αφήσουν τις χώρες τους εξαιτίας διώξεων, παραβιάσεων ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, κλπ. κλπ. Ότι οι τρίτες χώρες έτσι βρίσκονται κάτω υπό φοβερή πίεση και μιλάω και για ασφαλείς νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Μιλάω για ανθρωπιστικούς λόγους, για την εξέλιξη των εξωτερικών πολιτικών σε σχέση με τις ασφαλείς χώρες. Μιλάω για τη μεταχείριση των μεταναστών που επιστρέφονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία νομοθεσία για τα μεταναστευτικά ζητήματα, για τα δικαιώματα των μεταναστών ή τέλος πάντων ούτε καν για το δικαίωμα ασύλου και για την ανάγκη περισσότερο σήμερα από ποτέ κονδυλίων που να αφιερωθούν σε αυτό ακριβώ το θέμα. Συζήτησα κάπως με τους άντρους, αλλά ακόμα δεν τους έστειλα τροπολογίες για να συμπληρώσουμε την έκθεση αυτή, ακριβώς για να βάλουμε μια απόχρωση σε διάφορα ζητήματα και για να προσθέσουμε κυρίως ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι Σάντου συμφωνούν για το θέμα των απάτριδων. Και έχω και το θέμα των ευάλωτων προσώπων που ξέρω ότι θέλουν πολύ σκιώδεις εισηγητές. Επειδή ήξερα ότι έτσι καλλιώς συμφωνούσαμε γι' αυτό όλοι, το άφησα για τις τροπολογίες. Ότι πρέπει δηλαδή να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους, γυναίκες, παιδιά, και τους ε, πιο στο περιθώριο. Αυτά είχα εγώ να πω και από εκεί και πέρα περιμένω τα δικά σας σχόλια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να είμαι έτοιμη και εγώ με τις δικές μου τροπολογίες πριν υποβάλλετε εσείς τις δικές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Ο κύριος Ντεπρέ είναι ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ κύριε Ντεπρέ. Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο αντικαθαστώντας το Ερμήν Μισελ που είναι σκιώδης για το ζήτημα αυτό. Θα σας διαβάσω λοιπόν το κείμενο που ετοίμασε. Ναι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την κυρία Βερζιά για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Η έκθεση του Κοινοβουλίου έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει δήλωση της Νέας Υόρκης, αλλά και ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου που μας πέρασε, σχετικά με ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, είναι πολιτικά ε, σήματα ε, πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί το κοινοβούλιο μας. Η γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ πρέπει να αποτελεί προστεθέμενη αξία στην έκθεση. Θα ήθελα κυρίως να επιμείνω και πάλι στην ενίσχυση ε, και ανάκτηση νόμιμων και ασφαλών οδών. Είναι πολύ βασικό για την εξωτερική μας δράση στα θέματα της μετανάστευσης. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να, γίνει, να καταστεί πιο συγκεκριμένη στα πλαίσια των σχέσεών μας με τρίτες χώρες. Εξάλλου, η ανάκτηση των ασφαλών αυτών οδών θα πρέπει να γίνει και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα για την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Τέλος, σύντομα, άλλα στοιχεία, τα οποία είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, πιστεύω ότι πρέπει να προσταθούν στη γνωμοδότηση αυτή. Για παράδειγμα, η επιστροφή και πανεσδοχή το θέμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τους λαθροδιακινητές και την ε, εμπορία ανθρώπων, την εκμετάλλευση των ε, μεταναστών ουσιαστικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κριστίν Ρενόντε Μπονιφάη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, Μαρή Κριστίν Βερζιά αλλά και συγχαρητήρια. Γιατί το κείμενο αυτό με πλήρη τρόπο ακολουθεί τις διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας δράση για την μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις και με τις συστάσεις της νομοδότησής σου. Θέλουμε όντως να επικεντρωθούμε στις επιπτώσεις που έχει η πολιτική μας στα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων. Η πολιτική μας πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, κάτι το οποίο είναι ένα παραδιαγμάτευτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο αξιόπιστη εφόσον επίσης συνεργάζεται με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των πολιτικών μας για το εσωτερικό και το εξωτερικό, προκειμένου να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της ε, προσφυγιάς, να μην επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα της ε, ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων. Δεν πρέπει να επιστρέφουμε ανθρώπους σε χώρες όπου δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τους υποδεχτούν με ασφάλεια. Ζητάμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πεθύμησε και η συντάκτρια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να ανοίξει ασφαλείς οδούς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με διάφορους τρόπους, να υπάρξει ανθρωπιστική θεώρηση, να υπάρξει οικονομική ενίσχυση, μόρφωση, ε, πολιτική θεωρήσεων κλπ. Σε αυτά τα πλαίσια επιμένω κυρίως την ανάγκη εναρμόνισης σε προξενικό επίπεδο, κυρίως όταν πρόκειται για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Πρέπει επίσης να επιμείνουμε και σε άλλες πτυχές στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες, όπως είναι η πρόθεση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιδών δικαιωμάτων. Η εκπαίδευση, η μόρφωση, η απασχόληση, η βοήθεια στην ε, κοινωνική ένταξη είναι σημαντικά ζητήματα. Οι τροπολογίε μου θα πάνε προ την ίδια κατεύθυνση, όπω πάει και η γνωμοδότηση αυτή. Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στου πιο ευάλωτου, γυναίκε, παιδιά, αλλά και η ΛΟΑΔΑ. Υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βία μεγαλύτερος από τώρα που βρίσκονται σε εξορία. Άρα πρέπει να τους προστατεύσουμε και να έχουμε μία μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου όπως έγινε στην έκθεση που ψηφίσαμε την Άνοιξη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, στο οποίο θα επανέλθω με τις τροπολογίες μου, είναι η ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει δημοκρατικό έλεγχο όταν πρόκειται για συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, η νέα Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή πρέπει να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ για το κείμενό σου πάντως και είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βίντερ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Βλέπουμε μία κατάσταση όπου έχουμε 65 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς. Όχι βάζοντας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουν κοντά στους τόπους τους. Αυτή που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 65% οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι απορροφούν πόρους, ενέργεια που θα μπορούσαμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες. Στην πρόταση αυτή λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε, λέτε, ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοείται ε, ποσοστώσεις για τη μετανάστευση. Μα οι χώρες μέλη βλέπετε ότι δεν το κάνουν, ότι οι μισές χώρες δεν ακολουθούν τις συστάσεις για ποσοστώσεις για τους πρόσφυγες. Οπότε πώς θα γίνει αυτό. Να σκεφτούμε ανθρωπιστική βοήθεια στις τρίτες χώρες ίσως. Υπάρχει όριο για τον αριθμό των ανθρώπων μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έπειτα στην πρόταση δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την επιστροφή η Σουηδία. Να ξέρετε ότι πέρυσι πήρε πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που τελικά πρέπει να απομακρύνουμε, δεν θα μείνουν στη Σουηδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μας βοηθήσει για να τους επιστρέψουμε. Εμείς δεν έχουμε τους πόρους να το κάνουμε. 50.000 ανθρώπους πρέπει να απομακρύνουμε περίπου, αλλά δεν έχουμε τους σπόρους για να το κάνουμε αυτό. Πώς θα γίνει, πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Και έπειτα μια διευκρίνηση για τους εκτοπισμένους λόγω του κλίματος. Πώς θα διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Μαρή Κριστίν, λέει κυρία Πόστ, για τις προτάσεις της. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποιες συστάσεις, να προσταθούν στο κείμενο, αν συμφωνείτε. Στο σημείο 4, για παράδειγμα, θα ήθελα να το επεκτείνουμε λίγο και να πούμε μετά από τις ασφαλείς οδούς ε, κτλ. Να πούμε για να σταματήσει η λαθροδιακίνηση και η εμπορία ανθρώπων. Και στο σημείο 8 θέλω να προσθέσω ζητάει τη συλλογή ειδικών ε, δεδομένων και πιο πρόσφατων για τα δικαιώματα των ανθρώπων, κυρίως για τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και τους ΛΟΕΔ. στις χώρες προέλευσης εκείνων που ζητούν άσυλο, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών εκείνων που θεωρούνται ασφαλείς και μετά έχω και ένα 8α και μετά και ένα β όπου ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες που εργάζονται στις χώρες προέλευσης των ετούντων ε, άσυλο, ώστε να βρεθούν οι καλύτεροι δυνατόν τρόποι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και ομάδες ανθρώπων που είναι ευάλωτοι και το ΒΙΤΕΝ ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων των χωρών προέλευσης ώστε να βρεθεί ο καλύτερος μηχανισμός πρόληψης συγκρούσεων. Και εννοείται ότι θα συνεισφέρω και εγώ με τροπολογίες στο κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ιτζιν Λάμπερτ και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρή Κριστίν. Και συμφωνώ και εγώ με κάποια σημεία, κυρίως για τις νόμιμες οδούς. Και εγώ αμφισβητώ και την νομική βάση πολλών συμφωνιών εκείνη με την Τουρκία, με το Αφγανιστάν πιο πρόσφατα, όπου δεν είναι σαφές ποια είναι η νομική βάση για τέτοιες συμφωνίες και δεν έχει συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δε τεράστιες επιπτώσεις στις επιστροφές. Για τα θέματα της επανεισδοχής πρέπει να έχει λόγο το Κοινοβούλιο. Οπότε καλά κάνουμε και τα προσέχουμε όλα αυτά. Τώρα, γενικότερα, υπάρχει ανησυχία για το ότι επικεντρώνονται οι πολιτικές μας στο θέμα της μετανάστευσης και όχι της ανάπτυξης. Μα οι άνθρωποι που γίνονται μετανάστες ε, είναι ότι θέλουν να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προσόντα τους και τις δυνάμεις τους καλύτερα. Πάντως, πρέπει να μιλήσουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου. Αν ένας από τους στόχους μας είναι να μειώσουμε την ε, λαθροδιακίνηση ή όλες αυτές τις συμμορίες, θα πρέπει να εφαρμόζεται το κράτος δικαίου και στη χώρα προέλευσης. Είναι τα μέτρα που έχουμε μέχρι τώρα αποτελεσματικά. Το να παίρνουμε χρήματα από τέτοιες δραστηριότητες για να αποφύγουμε τη μετακίνηση των ανθρώπων είναι τελικά αντιπαραγωγικό. Τις ρίζες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε και τι επιπτώσεις έχουν οι επιστροφές σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα. Και το Πακιστάν που λέει ότι θα επιστρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο. Το Ιράν που θέλει επίση να επιστρέψει πρόσφυγες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει αποσταθεροποίηση το Αφγανιστάν. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Να είμαστε λοιπόν σίγουροι για το ότι αυτό που κάνουμε αποτελεί λύση για τη χώρα προέλευσης και όχι να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, αν έτσι το λέω κυρίως για το Αφγανιστάν, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε μετά για το πώς θα, προστα... πώς, θα προετοιμαστεί το Αφγανιστάν για να υποδεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αλλιώς είναι σαν να πετάμε τους ανθρώπους στη μέση της Καμπούλ και μετά δεχόμαστε να τους ευείτε οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό γιατί μερικές χώρες θέλουν να επιστρέψουν νέους, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχεδόν σχέση με τη χώρα προέλευσής τους, ούτε τη γλώσσα δεν γνωρίζουν καλά-καλά. Και νέοι άντρες. Εγώ καταλαβαίνω την ανησυχία μας για το ευάλωτες ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι τους νέους αυτούς άντρες πρέπει να τους ξεχνάμε. Και όσον αφορά την ασφαλή χώρα προέλευσης, το έχουμε συζητήσει πολύ νομικά. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι, για το ότι υπάρχει και μία διάσταση εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει την κάθε χώρα να την κρίνουμε, όχι βάσει τον στόχο μας στην εξωτερική πολιτική γενικά, αλλά βάσει του τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη χώρα. Μ' αρέσει που υπάρχει και η μία των ε, μεταναστών ε, λόγω κλίματος. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Να δούμε και πώς οργανώνουν οι διάφορες χώρες ε, το θέμα αυτό της μεταγκατάστασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Σίγουρα θα επανέλθουμε και θα καταλήξουμε σε κάτι, πιστεύω, ιδιαίτερα ικανοποιητικό για την Επιτροπή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, Τζιν. Η γνωμοδότηση αυτή έχει προκαλέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της συντάκτρια γνωμοδότησης και να καλωσορίσω και τους επισκέπτες που ήρθαν εδώ στην Επιτροπή μας. Η Νάταλη Κρίσπεκ τους έχει προσκαλέσει. Καλώς ήρθατε. Και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Θα έδινα το λόγο στην Μαρή Κριστίν. Όλο σε Γάλλους δίνω το λόγο. Δεν είναι ότι είναι Γαλλική Επιτροπή μας, μην νομίζετε. Αλλά πρέπει να δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δεν έχω τίποτα εναντίον τη. Μαρή Κριστίν, μου επιτρέπεις να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα ή θέλεις πρώτα εσύ να πάρεις το λόγο. Ωραία. Δύο λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να παρεύω από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποια σημεία που έθεσαν οι ευρωβουλευτές σας. για τις νόμιμες οδούς. Για τους μετανάστες και τους χρήζοντες προστασία. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο που μας πέρασε επέβαλε πρόταση για ένα πλαίσιο επανεγκατάστασης το οποίο συζητιέται μακροπρόθεσμα και προβλέπει ένα μόνιμο το οποίο ακριβώς να προσφέρει νόμιμες οδούς πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα τα οποία έχουν ε, ανάγκη από προστασία. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τις ευθύνες της και επιδεικνύει αλληλεγγύη απέναντι στους ε, υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο. και σε απελπισία. Τώρα για τις παρατηρήσεις που άκουσα για το κατά πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε ή όχι, για το πώς θα ενταχθούν και πάλι ε, στις χώρες όπου τους στέλνουμε. Για την Αφρική έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Έχουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα επιστροφών που περιλαμβάνει και την ένταξη των ανθρώπων αυτών στις κοινωνίες. Και θα έχουμε και άλλα τέτοια προγράμματα στο μέλλον με στόχο όχι μόνο να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν νόμιμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με ένα πακέτο επανένταξης που θέλουμε να είναι βιώσιμο, δηλαδή θέλουμε να έχει επιπτώσεις επιτόπου. Τέλος, για τις ανησυχίες που εκφράσατε για την τύχη που περιμένει τους ανθρώπους που στέλνουμε πίσω, υπάρχει η δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που λέει ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το σώμα. Μα το δείχνει και η έκθεση η οποία τακτικά δημοσιεύεται για την εφαρμογή της δήλωσης αυτής. Λέει η Τουρκία πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην Τουρκία να χαίρουν της αναγκαίας προστασίας. Θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι σύμφωνα με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου υπάρχει η εφαρμογή της έννοιας ασφαλής τρίτη χώρα. Εξετάζεται κατά περίπτωση η κάθε αίτηση ασύλου που επιτρέπει στη συνέχεια να καταλήξουμε στο κατά πόσο η τρίτη χώρα στην οποία θα επιστραφεί το άτομο θεωρείται ασφαλής για το συγκεκριμένο υποψήφιο επιστροφής. Κάθε υποψήφιος δηλαδή έχει δικαίωμα στη συνέχεια να αμφισβητήσει την έννοια αυτή της ασφαλούς τρίτης χώρας αν θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής. Και είναι ακριβώς αυτό που γίνεται στα hot spots στα ελληνικά νησιά όπου οι μετανάστες αυτοί που ζητούν διεθνή προστασία επικαλούνται το δικαίωμα αυτό το οποίο εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο στη Μαρή Κριστίν. Ναι, Άκουσα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά έκανα που περίμενα να μιλήσει εκείνη πρώτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε εδώ τους συναδέρφους, αλλά και συγγνώμη να ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ, τα λέω μα, έτσι, τα λέω από τα δόντια. Μας επαναλαμβάνεται μια ξύλινη γλώσσα. Δεν μας καθησυχάζετε. Εμείς θέτουμε κάποια ζητήματα. Το να μας μιλάτε νομικά δεν βοηθάει να καθησυχάσετε τις ανησυχίες που πολύ άριθμοι εδώ μέσα ε, συμμεριζόμαστε. Όταν ε, λοιπόν ακούω ότι καθημερινά ε, εφαρμόζουμε το μέτρο της επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας κτλ. δεν θα έχουμε συναντήσει τους ίδιους φαίνεται και δεν θα έχουμε διαβάσει και τις ίδιες εκθέσεις των ΜΚΟ που ανησυχούν για την κατάσταση. Άλλους θα έχετε δει εσείς, άλλους εμείς. Πάντως, εντάξει, ευχαριστώ τους συνεδέφου πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε, και αυτό είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο δεν έχω επιμείνει αρκετά, την ε, χειραγώγηση των στοιχείων. Γιατί πίσω από τα στοιχεία υπάρχουν πραγματικότητες. Ναι, 25.000 ε, εκτοπισμένοι και πρόσφυγες, αλλά από αυτούς το 65% εκατομμύρια. Συνεπώς πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να ξέρουμε τι σημαίνουν τα νούμερα αυτά στην πραγματικότητα. Υπάρχει βέβαια στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η Ευρωπαϊκή Ατζέντα πάντως που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα σημείο που αναφέρεται στις νόμιμες οδούς, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει αρκετά να γίνονται. Για τα τρία άλλα ναι, εντάξει, υπάρχουν κείμενα, όπως έλεγα και χτες πρόεδρε και εγώ δυσκολεύομαι να τα βγάλω πέρα γιατί πέφτουν το ένα μετά το άλλο με κάποιες διαφορετικές ε, οπτικές, αλλά εντάξει. Συνεπώς, η απάντηση, και αυτό λένε και οι σκιώδεις και όσοι πήρα το λόγο, η απάντηση νόμιμη οδή για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και επιμένω σε αυτό και μετανάστες και πρόσφυγες δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα πρόγραμμα μετακατάστασης. Η άφηξη πάντως στην Ευρώπη μειώνεται. Η οικονομική μετανάστευση μειώνεται. 1,7 εκατομμύρια ήταν, τώρα είναι 1,4 εκατομμύρια. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τις εκθέσεις των διάφορων σοβαρών οργανισμών, όπως είναι η Παγκοσμία Τράπεζα, το ΣΕΝΤΕ, όλοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνετε ανάποδα από αυτά που πρέπει να κάνει απέναντι στις προκλήσεις, τις δημογραφικές και οικονομικές που βρίσκονται μπροστά της. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν ακόμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης κάποια ανησυχία που αναφέρατε πολλοί από εσά. Το θέμα της κινητοποίησης όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της μετανάστευσης είναι ζωτική σημασία γιατί πράγματι βλέπουμε στην πράξη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο μένει στο περιθώριο των πολιτικών αυτών. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά εγώ σήμερα το πρωί διάβασα στις εφημερίδες ότι έγινε μια διάσκεψη υπουργών εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Δεν το ξέρω. Όταν οι Υπουργοί Εσωτερικών συνεδριάζουν, ε, θα έπρεπε και εμείς να ενημερωθούμε γιατί έχουμε και εμείς κάτι να πούμε από αυτού. Προσοχή λοιπόν. Είναι γνωμοδότηση ΛΥΜΠΕ, η ΑΦΕΤ παρακολουθεί στενά το ζήτημα, γι' αυτό εμείς να επικεντρωθούμε θα έλεγα στις τροπολογίες μας σε θέματα που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Για αυτά που καίνεται δικιά μας στην Επιτροπή Ακριβώς για να προσφέρουμε και εμείς μια προσθεθέμενη αξία. Νομίζω το κύριος ε, Ντεπρέ το είπε διαβάζοντας τα όσα του είπε ο συνάδελφος. Έτσι θα συνεισφέρουμε και εμείς στην έκθεση Αφέτ Ντεβε. Έχουμε πολλές ανησυχίες και συμμερίζομαι και τις ανησυχίες των συναδέλφων. Εύχομαι να συνεργαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Από τη Δευτέρα θα σας υποβάλω τις τροπολογίες μου για να μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε και με τους σκιώδεις και να έχουμε μια γνωμοδότηση μέσα στις προθεσμίες. Και που να είναι και καλή. Ευχαριστώ. Όλες και όλους. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου λοιπόν προθεσμία για να το γνωρίζετε και εσείς οι υπόλοιποι. Αναφερθήκατε στη συνάντηση με τους Αφρικανούς Υπουργούς Εσωτερικών, εννοείται αύριο, το, τους, ε, με, με, τις, χώρες ΑΚΕ. Όχι, δεν αναφέρεστε σε αυτό. Καλώς, καλώς. Δεν, θα παρατείνω τη συζήτηση, εννοείται κάτι άλλο. Καλώς. Όχι, δεν πρόκειται για τη συνάντηση με, τους, ε, με τις χώρες ΑΚΕ, αλλά πρόκειται για κάποια άλλη. Γιατί ορισμένοι υπουργοί έρχονται αύριο. Καλώς λοιπόν, ε, γι' αυτό σας ρώτησα, λέει ο Πρόεδρος. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα, σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους για την συζήτηση. Ας πάμε στα 24 και 25. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της εφισταμένης μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και της κρίσης ασφαλείας. Για το 2017 με σκιώδη Ισηγητή του Ματσόφσκι, επίσης και για τα δύο θέματα. Πρόκειται για σχέδια γνωμοδοτήσεων με προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών. Η κυρία Μακοβέη είναι εδώ. Δεν είναι. Α, φαίνεται πως έρχεται όμως η κυρία Μακοβέη. Να κάνω την εισαγωγή, θα έρθει στο μεταξύ, τι λέτε. Πέντε λεπτά. Θέλετε μια... Ε, θέλετε ένα διάλειμμα. Α, όχι, είναι επικίνδυνο, λέτε. Φαίνεται πως έχω βιαστεί ως τώρα. Uh, don't, don't take it personally. Don't... Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Mr. Dupre, a point of order to get some order into this meeting. Δεν θέλω να υπησέλθω στον ρόλο της κυρίας Μακοβέη, αλλά είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής Προπολογισμού. Αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η γνώμη μας. Απλό είναι. Τα λέω αυτά διότι έτσι θα μπορέσω να φύγω και νωρίτερα. Αλλά είμαι και σχεδόν συγητή τη ε, ομάδα των φιλελευθέρων. Πρόκειται λοιπόν για το δημοσιονομικό πλαίσιο που για 7 χρόνια βάζει την οροφή των εγκεκριμένων δαπανών στου διάφορου τίτλου του προπολογισμού. Ένα, δύο, ε, δύο α κτλ. Και για, τη, για τον τίτλο 3, εκεί η οροφή που εγκρίνεται, άνα βλέπω ότι προσέρχεται η κυρία Μα Κοβέη. Άρα όχι, θα τελειώσω, θα τελειώσω καλύτερα αντί να κλείσω το στόμα μου. Πρόκειται για τεχνικό θέμα. Αυτά που λέτε είναι ένα δημοσιονομικό ποίημα. Ε, ναι, λοιπόν, η οροφή αυτή είχε οριστεί σε μια εποχή που δεν αναμέναμε την ε, μεταναστευτική κρίση. Επειδή λοιπόν είναι καθορισμένη η οροφή και χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για να ξεπεραστεί η οροφή, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για να υπερβεί διεπηγούμε ε, την οροφή. Το ΔΕ Συμβούλιο Υπουργών ε, δεν επιθυμεί να αυξήσει την οροφή αυτή. Όμως, χάρη στην αποφασιστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί ευελιξίας και μάλιστα δύο. Ένας μηχανισμός ευελιξίας ή μέσο ευελιξίας για το contingency margin που επιτρέπει να κινητοποιηθούν κονδύλια και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές δεν είναι απόλυτα σαφές για τις προμές, είναι όμως για τις υποχρώσεις. Και αυτό που προτείνω εν προκειμένου είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών να υποστηρίξει με αποφασιστικότητα μάλιστα την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα δύο αυτά μέσα για να αυξηθούν τα συνολικά κονδύλια για τον τίτλο 3. ιδίω δηλαδή για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσεως και της μεταναστευτικής κρίσεως που αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω να υποστηρίξουν οι συνάδελφοί μου την έκθεση Μακοβέη. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα βρετανικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, αυξήσουμε τους, ε, ε, τα, τα ποσά. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι πρόκειται να υπάρξει κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις μεταναστευτικοί και άλλες που αντιμετωπίζουμε. Θα αναμείνω λοιπόν τη θαυμάσια έκθεση κυρίας Μακοβέη, την οποία υποστηρίζω και ζητώ από την Επιτροπή Λίμπε να, τα, να υποστηρίξει το περιεχόμενο της. Γεράρ, υπάρχει πολύ βρετανικό understatement στην Επιτροπή, μην ανησυχείτε. Ήθελα να πω ότι θαυμάσια τα είπατε και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μέλος στην Επιτροπή μας και έτσι υπάρχει και μια διασύνδεση με την Επιτροπή Προπολογισμών. Και από τα λόγια σα έμαθα και κάτι άλλο. Λοιπόν, έμαθα κάτι ακόμη. Και στο μεταξύ, βεβαίω, έχει προσέλθει η κυρία Μακοβέη. Αντιλήφθηνο ότι πρέπει να αποχωρήσετε. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σα. Μα βοηθήσατε πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Και εσεί τώρα, κυρία Μακοβέη. Μόλι μόλις κάναμε την εισαγωγή στο θέμα, σα παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο και να προχωρήσετε. Νομίζω ότι ακούσατε και τα τελευταία λόγια του Gérald Depré. Κοιτάξτε, θα μιλήσω ρουμανικά. Έτσι λοιπόν θα σας πω Instrumentul de flexibilitate ne asigură Μάλιστα, θα Πρόκειται για 130 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν ε, την δυνατότητα καθώς και την μέγιστη, τα μέγιστα ποσά που μπορούν να κινητοποιηθούν ε, αυτό το μέσο μέσα στο 2017 για να αντιμετωπιστούν οι επίγουσες ανάγκες. Έπειτα, τα επόμενα χρόνια, ακόμα και στην περίπτωση της δυνατότητας ε, κίνησης χρημάτων το τίτλο 3 ασφάλεια και πολίτες δεν θα είναι αυτά αρκετά τα χρήματα για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες. Αυτός ο προπολογισμό δεν είναι κατάλληλος. Η Κομισιόν θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσει από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα. Αυτά για τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του ε, προϋπολογισμού. Είναι το μέτρο το για την ευελιξία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά για τις δαπάνες για τις οποίες δημιουργήθηκε, για τις δαπάνες που είναι σαφώς ε, καθορισμένες και αυτές που δεν μπορούν να καλυφθούν από, άλλους, ε, από άλλα κονδύλια του προπολογισμού της Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει πολύ προσεκτικά να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή την πτυχή και αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Κατά δεύτερο λόγο, οι ανάγκες αυξάνονται συνέχεια στο πλαίσιο της κρίσης και κάνω έκκληση στην ε, υπευθυνότητα όλων όσον αφορά την κατανομή των ε, χρημάτων αυτών που πρέπει να διαιρεθούν με ισότιμο και διαφανή τρόπο ανάλογα με τις προτεραιότητες και να δαπανηθούν, όπως είπα, ξανά με διαφανή υπεύθυνο ε, τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμας είναι ο πρώτος σκιώδης που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ, που μου δίνει το λόγο. Απογοητεύομαι που βλέπω τόσους συναδέλφους που φεύγουν από αυτή τη συζήτηση, διότι δουλεύοντας για τον προϋπολογισμό, Ε, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Είναι σαν να, δουλεύει πάνω, να χορεύει κανείς πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Γιατί προσπαθείς να βρεις ε, τρόπους να λύσεις απρόβλεπτα προβλήματα, να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως αυτή που βρισκόμαστε τώρα στην Ευρώπη, όσον αφορά την μετανάστευση και την ασφάλεια. Η κρίση μεταναστευτική ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά εμείς σήμερα βλέπουμε τον αντίκτυπό της που είναι σαφής όσον αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό. Ο προπολογισμό του 2017 δεν είναι εξαίρεση από τις δύο προτάσεις της Κομισιόν για την κινητοποίηση της, του μέσου ευελιξίας ώστε να χρηματοδοτηθούν τα προβλήματα της ε, κρίσης μετανάστευσης και επίσης να χρησιμοποιηθεί το περιθώριο που υπάρχει. Εμείς υποστηρίζουμε αυτήν ε, την πρόταση ο ΕΛΚ. Και, Όσον αφορά την πρόταση του κ. Ντεπρέ, τη στηρίζουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ευελιξίας. Ε, έχουμε τώρα της τους τίτλους 2 και 5 και χρειάζεται να, το να τους χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες καταστάσεις στην Ένωση. Γιατί στην 3 έχουμε φτάσει στο μάξιμο, έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο. Οπότε, χωρίς το μέσο ευελιξίας, δεν θα μπορέσουμε καν να χρηματοδοτήσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε επί τη βάση της ε, κρίσης της μετανάστευσης. Η Κομισιόν έκανε πρόταση και για τις, ε, την ακτοφυλακή και για τη συνοριοφυλακή. Και χωρίς επιπλέον χρήματα αυτά θα μείνουν ε, μόνο στο χαρτί. θα είναι κάτι που θα μπορεί να λειτουργήσει μόνο στην εικονική πραγματικότητα και όχι στον πραγματικό κόσμο. Τέλος, αυτά τα χρήματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επόμενα χρόνια και όταν θα αναθεωρήσουμε το PDP θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μπούμε πάλι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση. Για την συνάδελφο Μακοβέη έχω δύο μηνύματα από το ΕΛΚ. Η πρόταση είναι αρκετά τεχνική, αλλά πάλι πρέπει να αναφέρω δύο προτεραιότητες ε, του ΕΛΚΑ που τις επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια. Θέλω λοιπόν να πω ότι η πρόταση της συναδέλφου Μακοβέη είναι πολύ καλά ισορροπημένη έχει την υποστήριξή μας, αλλά υπάρχουν δύο σχόλια που έχουμε να κάνουμε, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για Europol, η Europol πρέπει να ενισχυθεί και καθώς επίσης οι νεοσυσταθήσεις ε, ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Επίσης, τι θα γίνει με την χρηματοδότηση της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Και η δεύτερη παρατήρηση ε, είναι η δίκαιη κατανομή των οικονομικών προτεραιοτήτων. Ε, αναφέρθηκε και από τη Μόνικα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε διαφάνεια, λογοδοσία και λογική χρηματοδότηση, σοφή χρηματοδότηση. Είπα το ίδιο και στην ε, συνεδρίαση της ΚΟΝΤ. Είναι πολύ σημαντικό η χρήση όλων των δημοσιονομικών μέσων να είναι διαφανής ή εν πάση περιπτώσει πιο διαφανής. Είναι αδύνατο να αγοράζουμε πράγματα τελευταία στιγμή και τελευταία, μάλλον να, να, να, πληρώνουμε για πράγματα για τελευταία στιγμή, ε, γιατί δεν έχουμε κάνει σωστά τη μοιρασιά για ένα μακροχρόνιο διάστημα. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε βραχυπρόθεσμα προβλήματα, ξαφνικά πρέπει δηλαδή να κινητοποιηθούν τα κονδύλια αυτά άμεσα, ε, να καλυφθούν projects και αυτό πρέπει να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Το έχεις ήδη παρατηρήσει ότι πρέπει ε, όντως να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Ήθελα ε, και εγώ να το τονίσω. Έχει το λόγο, Μπεργκίτε, που αντικαθιστάσε τον ε, σκιώδη του των σοσιαλιστών. Ο Ντανιέλ δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ το πρωί. Ε, Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότηση και από απλά τεχνικά, από, τεχνική άποψη οι σοσιαλιστέ δεν έχουν να κάνουν σοβαρά σχόλια. Ε, ε καλωσορίζουμε την ε, αύξηση του τίτλου 3 στο σχέδιο προϋπολογισμού της ε, Κομισιόν και είναι καλά νέα ότι η πρόταση για τη χρήση στο maximum αυτής της, ε, αυτού του περιθωρίου είναι θετική. Ε, αυτό θα εξασφαλίσει απάντηση στην πρόκληση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης για το 2017. Θα μείνουν οι δυνατότητές μας στο ίδιο επίπεδο με το 2016. Ωστόσο το μέσο ευελιξίας ε, δεν αρκεί ούτε το περιθώριο αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες στη τίτλο 3 γιατί δεν αναμένεται να μειωθούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες το 2017 και τα κράτη μελη που είναι στην πρώτη γραμμή θα παραμείνουν υπό μεγάλη πίεση. Η αναθεώρηση του PDP, όπως παρουσιάζεται από την Κομισιόν, προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση ε, 2,550 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μπαίνουν για την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή και 5,5 δις για την μετανάστευση. Η άφηξη μεταναστών δεν θα πρόκειται να σταματήσει στο εγγύς μέλλον και γι' αυτό και θα πρέπει αυτή η, η, η περίοδος να είναι ευέλικτη. Ελπίζουμε ότι το επόμενο PDP θα το αντικατοπτρίσει αυτό με τα κατάλληλα μέσα ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει συνεχιζόμενη πολιτική κρίση ασφάλειας και κρίση προσφυγική. Είναι μια πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση και ε, είναι σωστό να λυθούν τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα στα με τρόπο. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Πριν να στραφώ στην εισηγήτρια. Α, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια και να Δεχτώ την ε, πρόταση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν, να κινητοποιηθούν τα δύο μέσα ευελιξίας και το κινητό περιθώριο για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ε, ταυτόχρονα και αυτό θα αντικατοπτριστεί και στις ε, τροπολογίες που θα καταθέσω. Πιστεύω πως η χρηματοδότηση της Ένωσης για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών και των ετωτών θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη σε αντιπαράθεση με τις ε, απόλυτη, την απόλυτη προτεραιότητα που δίνεται τώρα στην ε, έλεγχο της ασφάλειας και τα μέτρα της ασφάλειας Πολύ αφισβητήσιμα είναι όλα αυτά τα μέτρα από την άποψη της δημόσιας ηθικής όσον αφορά τη διοικητική κράτηση. Ε, μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχουν δείξει να είναι αποτελεσματικά και που πολύ συχνά ε, παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών. Ή, τροπο, στις τροπολογίες μου σκοπεύω λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή να χορηγήσει επιπλέον πόρους κατά προτεραιότητα στις δράσεις που έχουν απευθύνονται στα κάτι μελη που αναλαμβάνουν δράσεις που στόχο έχουν την υποδοχή. Και κυρίως, δεδομένου ότι θεωρώ πως είναι επίγον να βγούμε από τη λογική της επίγουσας κατάστασης και να μπούμε στη λογική διαρθρωμένων μέτρων, και δράσεων λοιπόν που θα έχουν στόχο να ενταχθούν οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Ε, θα τα υποβάλω όλα αυτά με τις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και στρέφομαι και πάλι στην κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συμβολή τους και... Περνάμε και στο επόμενο. Θα, θα, μάλλον θα σας πω ότι θα λάβω υπόψη όλες σας τις απόψεις ε, στην ε, ε, ολοκλήρωση, μάλλον στην ε, Τελική επεξεργασία. Μάλιστα, προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 30... 21η με του Οκτωβρίου. Πάμε στο σημείο 26, ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τις σχετικές βάσεις δεδομένων. Και η συγκήτρια θα μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στις 11 Οκτωβρίου. Εισαγωγικά να σας πω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτός ο φάκελος ανήκει σε ένα πακέτο προτάσεων της Κομισιόν που έχει ε, στόχο την ανείχνευση τρομοκρατών της ε, ώστε να εμποδιστούν να κάνουν επιθέσεις. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Έχετε το λόγο για να μας πείτε πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. A uh, Σας ευχαριστώ. Εξήγησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας ότι αυτή η πρόταση είναι στοχευμένη ειδικά στην αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη κυρίως λόγω του φαινομένου των ξένων μαχητών. Η σημερινή πρόταση επιτρέπει να εντοπιστούν οι κάτοικοι Ευρωπαίοι πολίτες που είναι μέλη του ΝΤΑΕΣ και που ε, επιτρέπει στα κρατημέλη να, κάνουν, να προβαίνουν σε συστηματικούς ελέγχους όπως στην ε, διαβούλευση των ε, βάσεων δεδομένων πάνω απ' όλα του ΣΥΣ για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες και μη Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που έχουν περάσει τα εξωτερικά μας σύνορα. Συμφωνούμε όλοι για το γεγονός ότι η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε συμφωνία σε σχέση με αυτήν την ε, έκθεση, ακόμα και αν έχει υποβληθεί από το 14 από την Κομισιόν εχθές. Στη... Υπήρξε ένα τριμερής, αλλάζουν κάπως οι προτάσεις, ελπίζω πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η συζήτηση στον τριμερή. Υπάρχουν ε, δύο επίμαχα πολύ ζητήματα, ένα είναι τα αίτια για την εξαίρεση από τον κανόνα συστηματικών ελέγχων και για την εφαρμογή, την διενέργηση μάλλον ε, στοχευμένων ελέγχων. Η εξαίρεση μπορεί να υπάρχει μόνο στην περίπτωση όπου ένα όπου το σύστημα είναι δυσανάλογο και επηρεάζει τη ροή του κυκλοφορία. Το Συμβούλιο την υποστηρίζει αυτή την ε, πρόταση και ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να ανατρέχουν σε στοχευμένου ε, ελέγχους από τη στιγμή που θεωρούν πω οι συστηματικοί αυτοί οι έλεγχοι έχουν ε, δυσανάλογο αντίκτυπο για πολλούς και διάφορου λόγου. Υπάρχει ένα ανοιχτό κατάλογο στο δεύτερο επίμαχο θέμα και σχετίζεται με το πρώτο και αφορά το είδο των συνόρων όπου μπορεί να διενεργούνται αυτοί οι στοχευμένοι έλεγχοι ως εξαίρεση από το γενικό κανόνα. Η πρόταση αναφέρεται σε αυτά τα χερσαία μόνο και θαλάσσια σύνορα και το Συμβούλιο συμφωνεί διότι λέει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και για τα εναέρια σύνορα. Υπάρχει ήδη υποδομή για να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σε πολλά ε, αεροδρόμια και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Λίμπε ενέκριναν κείμενο που επιτρέπει την ίδια μεταχείριση για όλα τα είδη συνόρων. Δηλαδή να γίνονται εξαιρέσεις και στα αεροδρόμια. Τα σημεία αυτά είναι ακόμα ανοιχτά Πρέπει ακόμα να συζητηθούν. Η θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι διαφορετικές. Όπως είπα, στον χτεσινό ε, τριμερή έλαβα μια συμβιβαστική από πλευρά του Συμβουλίου για μια μεταβατική περίοδο 9 μηνών για τα ε, ε, αεροδρόμια, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και στη συνέχεια θα, γίνουν, θα γίνονται συστηματικές, συστηματικοί έλεγχοι και στα σύνορα των αεροδρομίων. Τώρα, με το Συμβούλιο βρήκαμε μία λύση σε ένα άλλο επίμαχο θέμα, βάσει δεδομένων Τα κράτη-μέλη, είπαμε, θα πρέπει να δίνουν πλήρης και ε, ε σωστές πληροφορίες ε, άμεσα προς το ΣΥΣ. Ε, αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι η πρώτη με την οποία ερχόμαστε σε διαβούλευση. Δηλαδή δεν αποκλείει άλλες βάσεις δεδομένων, ούτε διεθνεί βάσεις, αλλά με την προϋπόθεση ότι το ΣΥΣ θα τροφοδοτείται με τις πληροφορίες που πρέπει. Κοντεύουμε λοιπόν εδώ να φτάσουμε σε συμφωνία, που ελπίζω ότι θα μας οδηγήσει και στην ολοκλήρωση του κειμένου. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ε, συμφωνία και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε πριν το τέλος του έτους. Θα υπάρξει επόμενο τριμερής ε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Μακοβή. Έχω που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο. Είναι πραγματικά δραματικό το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν αυτά. ...170 πολίτες ζεστάλησαν πίσω από τη Γερμανία στη Συρία μέσα σε ένα μήνα, τον προηγούμενο μήνα. Πράγματι είναι δραματικό το πλαίσιο. και το θέμα βέβαια είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο και αυτά που γράφεται είναι πολύ λεπτομερή. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις. Η Μπάρμπαρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων φαίνεται να σημειώνεται κάποια πρόοδος, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται να αναζητηθεί μια συνένεση και μάλιστα ως το δυνατόν συντομότερο. Πρώτα-πρώτα μας απασχολεί η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ελπίζω και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες και ιδίω των σοσιαλιστών και δημοκρατών θα μπορέσουν να συνενέσουν μαζί μας ώστε να προχωρήσουμε ταχύτερα. διαπραγματευόμαστε το σχέδιο εδώ και ένα εννεάμινο, δηλαδή πολύ καιρό. Για το Λαϊκό Κόμμα ο στόχος είναι να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση που να επιτρέψει στον κανονισμό να τεθεί σε εφαρμογή σύντομα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Σοφή Ιντφέλτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση. Συμφωνώ με την προσέγγιση της, δηλαδή να εντοπιστούν κάποια στρατηγικά θέματα πριν αρχίσει ο τριμερής διάλογος για να γνωρίζουμε ποια πράγματα είναι σημαντικά για μας και πού ενδεχομένως υπάρχει περιθώριο λιγμών. Τονίστηκε ότι το θέμα θεωρείται κατεπήγον. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραιτηθεί από την θέση του. Γνωρίζω ότι το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα άκαμπτο. Εάν το θέμα όμως είναι ε, κατεπήγον, αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλες οι πλευρές να δείξουν κάποια ευκαμψία. Έχω δε την αίσθηση ότι εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε τα τέσσερα σημεία, δηλαδή ίση μεταχείριση όλων των ειδών συνόρων το ερώτημα υπό ποιες συνθήκες μπορούν να αντικατασταθούν η συστηματική έλεγχοι από δειγματοληπτικούς πρόσβαση σε ποιες τράπεζες δεδομένων. Και, τέλος, και τέλος η καταληκτική ρήτρα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ υποφώσκουν κάποια θέματα που δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι χώρες μέλη χρησιμοποιούν το ΣΥΣ και διοχετεύουν σε αυτό τις πληροφορίες και ιδίως μετά από τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Ακούμε άλλα πράγματα βέβαια τώρα. Τότε όμως είχαμε δει ή είχε διαπιστωθεί ότι δεν διοχετεύουν επαρκή δεδομένα οι χώρες μέλη στο ΣΥΣ. Έχουμε και την κάπως άκαμπτη στάση του Συμβουλίου που οδηγείται από την επιθυμία ορισμένων χώρων μελών να πιέσουν άλλες που προφανώς δεν συνεργάζονται. Αλλά αυτό δεν είναι η δική μας δουλειά. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να πούν μάλιστα αναμένουμε από εσά να χρησιμοποιείτε το ΣΥΣ και να διευθετεύετε τις ε, δεδομένων στο σύστημα αυτό. Δεν γίνονται αυτά σε τριμερείς διαλόγους. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών αλλά ταυτόχρονα να τηρούνται και οι θεσμικές μας αρχές. Γιατί εγώ έχω ακόμη μεγάλα ερωτηματικά σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας, όχι ταυτοτήτων, έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να γίνονται συστηματικά. Και πώς αυτό συμβαδίζει με την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και της επικουρικότητας. Διότι μειώνουμε και δραματικά μάλιστα την ελευθερία των χωρών μελών να προβαίνουν σε ίδιες επιλογές. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω πάντως ότι θα διεξαχθεί σύντομα άλλο τριμερής διάλογος που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε μια λύση στη βάση των γραμμών που πρεσβεύει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Μόνικα Χολμάιερ. Ορίστε. στη βάση της αναλύσεως που έκανε η Σοφή κάπως εκπλήσωμε διότι όταν βλέπω τα πράγματα, εγώ τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι οι χώρες μέλη για την ώρα έχουν λάβει σωστές αποφάσεις. Εμείς οι ίδιοι είπαμε μάλιστα ότι θέλουμε ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Να γνωρίζουμε ότι όποιος εισέρχεται στην επικράτεια πρέπει να είναι γνωστός. Δεν, χρειά, δεν, θα, πρέπει δηλαδή να χρειάζεται να εξηγούμε στους πολίτες μας γιατί εγκληματίε, τρομοκράτε και ούτω καθεξής οι οποίοι μάλιστα διέρχονται σύνορα καμιά φορά και με το πραγματικό του όνομα, γιατί τελικώ δεν συλλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν, εφόσον γίνονται έλεγχοι, για παράδειγμα στα αεροδρόμια, θα πρέπει να πω με νυφάλιο τρόπο. Ο, στο αεροδρόμιο απαιτείται συστηματικός έλεγχος. Δεν μπορώ να πω στο αεροδρόμιο, ε, κάπου κάπου αφήνω και κανέναν. Ωραία, αφήνουμε τότε τους επόμενους πέντε και τους επόμενους 100 και μετά ε, απορχίζω ξανά. Γνωρίζουμε και για τα χερσαία σύνορα, για παράδειγμα στο Γιβραλτάρ, όπου η κυκλοφορία εκεί είναι τεράστια και επειδή είναι εξωτερικά σύνορα γίνεται συστηματικός έλεγχος και από τις αρχές του Γιβραλτάρ χωρίς να ανακόπτεται ωστόσο η ροή της κυκλοφορίας. Δεν θέλουμε βεβαίω φορτικά αυτοκίνητα να παραμένουν μπροστά από τα σύνορα, δηλαδή ε, ε, να μην μπορούν να διέλθουν τα σύνορα ασφαλώς. Όχι, δεν θέλουμε να υποστεί μία η οικονομία. Θέλουμε όμως να χρησιμοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι που να επιτρέπουν την διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων. Ναι, εγώ επιθυμώ και στα εσωτερικά σύνορα να μπορέσουμε να άρουμε το δυνατόν συντομότερο τους ελέγχους. Δεν θέλουμε να έχουμε σε κάθε εσωτερικό σύνορο, μεταξύ χωρών μελών δηλαδή, να έχουμε ελέγχου και μάλιστα ακόμα λιγότερο συστηματικού ελέγχου. Επειδή όμω τα σύνορα, ε, συγγνώμη, επειδή τα αεροδρόμια πάντοτε είναι στην ουσία εξωτερικά σύνορα αφού δέχονται διεθνεί πτήσει και τα αεροδρόμια του ή άλλω είναι ιδιαίτερα ευαίσθητε ζώνε, θα πρέπει να γίνονται συστηματικέ. ελέγχοι. Και τελευταία υπόθεση που ε, διαρευκάνθηκε στην Γερμανία, ε, ε υπόθεση δηλαδή ε, προπαρασκευαστικής τρομοκρατικής επιθέσεως, πάλι θα στρεφόταν κατά αεροδρομίου. Το Συμβούλιο δεν είναι άκαμπτο, αλλά πρέπει στο κάτω της γραφής να αντιμετωπίσουμε και λίγο τι λέει ο κόσμος. Κανένας δεν κατανοεί πώς αφήνουμε να περνούν τρομοκράτες από τα εξωτερικά σύνορα, είτε διότι δεν ελέγχεται το Eurodac, και εδώ δεν έχει σχέση με τη δική σου ερώτηση βεβαίως, αλλά και στα εξωτερικά σύνορα δεν διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι. Με τον τρόπο όμως αυτό επιτρέπουμε να αυξάνεται η εσωτερική δυσπιστία των πολιτών και αυτό αφήνει χώρο σε λαϊκιστές οι οποίοι έρχονται και λένε βεβαίως σύνορα διότι αυτά θα καταστήσουν ασφαλή την Ευρώπη και επομένως και εσωτερικά σύνορα και φραγμοί κλπ. Εγώ θέλω το Σέγγεν να μπορέσει να, να, να, λειτουργήσει και πάλι, να ξεχάσουμε τα εσωτερικά σύνορα, να μπορούμε να εμπιστευόμαστε εμένοι τους δε. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνονται στα εξωτερικά σύνορα οι έλεγχοι. Και αυτό σημαίνει επίση ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Το να μην επιτρέπουμε συστηματικού ελέγχου στα αεροδρόμια, για μένα μου φαίνεται ότι αυτό ανοίγει τι πόρτε σε μεγάλο κίνδυνο. Και πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Ας μην αρχίσουμε τώρα στη διαπροσωπική συζήτηση. Σοφή Ιντφέλτ. Παρακολουθούν ίσω ε, πολίτε τη συνάντησή μα και θα ανησυχούν πολύ από αυτά που άκουσαν. Εγώ θέλω λοιπόν να πω Ωραία, μία διευκρίνηση σύντομα. Μα αφήνετε να μιλήσω. Τι λέτε τώρα, λέει η κυρία Ιντφέλτ. Διευκρίνηση. Διαπραγματευόμαστε στην βάση τη θέσεω που έχει ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμβασμό. Δηλαδή δεν ικανοποιεί ούτε εσά ούτε εμένα απολύτω. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συστηματικών σε σύγκριση με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Δεν λέμε ότι τα αεροδρόμια αποφασίζουν με το έτσι θέλω να κάνουν απόκληση, να έχουν εξαίρεση δηλαδή από του συστηματικού ελέγχου. Η μόνη εξαίρεση στην οποία συμφωνεί άλλωστε και το Συμβούλιο είναι μια εξαίρεση που δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια, παρά μόνο με τι ροέ τη κυκλοφορία που δεν έχει καμιά έννοια. Αυτό που θέλουμε εμεί είναι να υπάρξει μια εξαίρεση στη βάση αξιολόγηση του κινδύνου και στη βάση κοινών δικτών. Αυτά έχουν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Και δεύτερο, εάν ανησυχούμε, και αυτό είναι που με ενοχλεί πολύ, Όλοι ανησυχούν για την ασφάλεια. Κυρία Χολμάιρ, να ακούστε τι λέω. Εάν όμως οι χώρες μέλη ανησυχούσαν το ίδιο για την ασφάλεια όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπραταν το καθήκον τους και θα γέμιζαν με δεδομένα το SIS. Θα φρόντιζε δηλαδή το SIS, το Schengen Information System, να είναι πλήρες. Δεν το κάνουν όμως οι χώρες μέλη και προσπαθούν τώρα μέσω των διαπραγματεύσεων αυτών να πιέσουν οι μέλη δε. Ναι, αρχίσατε τελικώ διάλογο. Τώρα θα χρειαστεί να δώσω και πάλι τον λόγο στην κυρία Χολμάιρ για να απαντήσει. Αλλά παρακαλώ σύντομα. Και μετά να ακούσουμε την κυρία Μακοβέη πάλι. Θα είμαι σύντομη. Δεν μπορούμε να επανερχόμεθα συνεχώς στα παλιά. Οι χώρες μέλη το έχουν κατανοήσει πλέον ότι πρέπει να τροφοδοτούν το SIS. Το κατανόησαν αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να επανερχόμεθα στα ίδια και στα ίδια. Αυτό όμω δεν σημαίνει, δεν αποτελεί δικαιολογία για ποιον λόγο να μην γίνονται συστηματικά έλεγχοι. Διότι στα τα αεροδρόμια δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γνωρίζει ποιο τρομοκράτη θα επιλέξει ποιο αεροδρόμιο για να προσπαθήσει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αρκετά ευφυεί και τρομοκράτε για να αντιληφθούν και αυτοί την ε, ε, αξιολόγηση των κινδύνων. Έχουν μάλιστα θαυμάσει connections, μην ανησυχείτε καθόλου. Κυρία Μάκοβη, σα παρακαλώ να κάνετε μια σύνοψη και μάλιστα σύντομα. Πρόκειται για έκθεση για τριμερή διάλογο. Μια φράση σας παρακαλώ κυρία Μακοβή. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Δεν έχει μικρόφωνο κυρία Μακοβή. συνεχίζει ο πρόεδρος. Ε, έχετε στην ουσία ήδη ε, εξαγάγει τα συμπεράσματα σας. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στις επόμενες διαπραγματεύσεις, στις ημερούς διαλόγους. Σας ευχαριστούμε πολύ και όλοι. Νομίζω τελειώσαμε κιόλας. Τι άλλο μείνει. Όχι, ε, Συνεχίστε λοιπόν, μια και δεν βρήκε ακόμη το, το επόμενο θέμα τη ημερησίας διατάξεω. Η κυρία Μακοβέη, στα αγγλικά, περιμένουμε πληροφορίες από την Εουλίσα. Α, τελειώνουμε, την This is the end, κυρία Μακοβέη. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λέει η κυρία Μακοβέη. Για την προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ζωτική σημασία την ατζέντα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Συμφωνώ με τη Μόνικα, δεν μπορούμε να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε να μας ξανακτυπήσουν μόνο και μόνο επειδή κάποιες χώρες μέλη δεν, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους. Έχουν αρχίσει τώρα, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, πολύ περισσότερες χώρες τροφοδοτούν ε, τα δεδομένα της Europol. Το λάθος μου, λέει ο Πρόεδρος, είναι ότι κάθε φορά ρωτώ πολιτικούς εάν πραγματικά θέλουν να μιλήσουν. Ε, είναι προφανής η απάντησή τους, έτσι είναι. Εγώ αυτή λοιπόν. Α, έχουμε τα διάφορα τώρα. Υπάρχει κανένα διάφορο, δεν υπάρχει κανένα διάφορο. Επόμενη συνάντηση. Νομίζω ότι όντω ε, ε, ήταν ισορροπημένε οι παρεμβάσεις. Στις 17 Οκτωβρίου στι 3 το απόγευμα. η συνεδρίαση.